Good morning everybody. Καλημέρα σας. Μπορείτε να κάνετε δεκτή την ημερήσια διάταξη σήμερα και όχι αύριο. Σας θυμίζω ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο ζωντανή συνεδρίαση. θα έχουμε κάποια ένα σεμινάριο γύρω από τα θέματα αυτά. Για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ηλεκτρονικά γύρω από τη συνεδρίασή μας, τα λεγόμενα e-meeting. Έχουμε επίσης και το δελτίο της Επιτροπής μας, το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει τώρα για τις ακροάσεις. Εμείς θα τις συζητήσουμε στα πλαίσια των συντονιστών σήμερα το απόγευμα. Αλλά η επόμενη πέμπτη είναι μια δύσκολη μέρα για μας, για την Επιτροπή μας. Είμαστε η δεύτερη Επιτροπή στην Ακρόαση Μοσκοβίτσι. Έχουμε επίσης και την Ακρόαση Βεστάγγε μέχρι αργά το απόγευμα. θα πρέπει μετά από κάθε ακρόαση να συναντώνται οι συντονιστές και να παίρνουν αποφάσεις για το τι συνέχεια ε, θέλουν να δώσουν, να στείλουν μια επιστολή στήριξης ή όχι. Εγώ θα συζητήσω τα θέματα αυτά με τους υπόλοιπους Προέδρους Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Κάποιες από τις προτάσεις πάντως που έχουμε πάρει μέχρι τώρα ίσως να καταστήσουν δύσκολη τη μετακίνησή σας την πέμπτη του απόγευμα και υποπτεύομαι ότι θέλετε να φύγετε την πέμπτη του απόγευμα και γι' αυτό θα προσπαθήσω να το πετύχω αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θα μαζέψω περισσότερες πληροφορίες τις οποίες θα μεταφέρω στους συντονιστές σήμερα το απόγευμα. Λοιπόν, ε, εντάξει τα πρακτικά γίνονται δεκτά. Ας περάσουμε τώρα στο βασικό θέμα για σήμερα. Να σας παρουσιάσω τον συνάδελφο, διευθυντή της τρίτης διεύθυνσης για την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Θα μας μιλήσει για την έκθεση για το κόστος της μη Ευρώπης, το οποίο σας απασχολεί εδώ και αρκετούς μήνες. Ήταν τμήμα των αναγνωσμάτων μου το καλοκαίρι άλλωστε και θα μας φέρει σε επαφή και με τους εμπειρογνώμονες που παρουσίασαν τα πέντε διαφορετικά κομμάτια της έκθεσης αυτής. Καθένας από εσά γύρω στα πέντε λεπτά και μετά ερωτήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε τις πρώτες τρεις παρουσιάσεις και μετά θα αρχίσουν οι ερωτήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, σε ερωτήσεων μετά από τις τρεις πρώτες ομιλίες και μετά οι επόμενες. Και μετά πάλι ερωτήσεις. Και θα μας πείτε πότε θα είναι διαθέσιμο και στις υπόλοιπες γλώσσες το κείμενό σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι χαρά που βρίσκομαι στην ΙΜΚΟ, λέει ο κύριος Ντάν. Επειδή έχω εργαστεί για αρκετά χρόνια στην Επιτροπή σας, γνωρίζω το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σήμερα το πρωί πάντως εκπροσωπώ τη Διεύθυνση για τη μελέτη των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας που δημιουργήθηκε το 2012 από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου για να δώσει ακριβώς στο Κοινοβούλιο νέα μέσα ελέγχου και να καταστήσει το Κοινοβούλιο ικανό να κάνει ε, μελέτες επιπτώσεων ε, πιο αποτελεσματικές από ό,τι σήμερα. Σήμερα το πρωί έχουμε λοιπόν την ε, πρόταση αυτή, το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε, βλέπετε ότι είναι ένα μεγάλο κείμενο και σίγουρα μπορούμε να μεταφράσουμε τα συνθετικά κείμενα σε όλες τις γλώσσες και εφόσον ζητηθούν περισσότερες λεπτομέρειες οι επιμέρους μελέτες μπορούν να μεταφραστούν και αυτές. Αυτό είναι ελέγξιμο βέβαια. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε διατεθειμένοι να σας δώσουμε το υλικό το οποίο θεωρούμε και εμείς ότι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο σε επίπεδο επικοινωνίας για το Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μία επιστροφή στα βασικά. Δηλαδή δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αυτό που γέννησε τον όρο, τη φράση ε, κόστος της μη Ευρώπης από το 1993, ε, Άλμπερτ και άλλων τότε ακριβώς είχε, είχαν συλλάβει την ιδέα ότι υπάρχει κόστος για την έλλειψη της Ευρώπης και ο καθηγητής Τσεκίνη με τη μελέτη του το 1998 εξετίμησε ότι το κέρδος για την ενιαία αγορά ήταν 200 δις εκεί, όπως ε, ε, το λέγαμε τότε. Ε, αυτό σημαίνει σήμερα 800 περίπου δις ευρώ. Αυτό που μας ζητήσατε να κάνουμε δηλαδή είναι εμείς να ενημερώσουμε λίγο την έκθεση τσεκίνη. Εντοπίσατε πέντε τομείς στους οποίους σου ζητήσατε επιμέρους πληροφορίες και πέντε εμπειρογνώμονες κατέθεσαν τις μελέτες τους στους τομείς αυτούς. Εσείς ξέρετε σε ποιους θα δώσετε το λόγο, αλλά νομίζω ότι ακριβώς κάλυψαν τους τομείς αυτούς και αυτό μας επέτρεψε να προχωρήσουμε. Οι εμπειρογνώμονες δούλεψαν ανεξάρτητα, δεν συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Έχουμε λοιπόν πέντε εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους απόψεις για την ενιαία αγορά. Συνοπτικά τώρα, ίσως είναι δύσκολο να διαβάσετε τους πίνακες που έχετε μπροστά σας. Ο Χάφνερ θα μας μιλήσει για την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών. Εκεί βλέπετε ότι υπάρχει ε, ε, το κατώτερο είναι 183 δις κατέτος. Ε, μετά θα μιλήσουμε για την ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών. 338 δις είναι η εκτίμηση. Ο Μέιτ θα μας μιλήσει για τις δημόσιες προμήθειες. 36 δις. Ο Μπρεζίνσκι θα μας μιλήσει για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχουν δύο μελέτες εδώ και η μελέτη για το κεκτημένο για τους καταναλωτές, η μία 36 δις και η άλλη 58 δις κατέτος. Νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ υψηλά ποσά βέβαια και μπορεί κανείς ε, να προσθέσει και τις εκθέσεις τις οποίες πρόσφατα έχουμε και έχει κυκλοφορήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφαιρώντας τα επικαλυπτόμενα μπορούμε να υπολογίσουμε ότι συνολικά μιλάμε για οικονομικά κέρδη 632 δις. Συνολικά μπορούμε να φτάσουμε σε μακροπρόθεσμη λογική 1,33. Ε, μιλάμε για τρομακτικά ποσά σημαντικού, μεγάλη σημασίας και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό αναπτυξιακό. Εγώ στις συνθετικές εκθέσεις ε, έχω συμπεριλάβει και κάποια πρώτα συμπεράσματα, τα οποία είναι προσυζήτηση βέβαια. Τα συμπεράσματα αυτά αναφέρονται στο ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δυσκολίας είναι ότι υπάρχει ένα διακανονιστικό πλαίσιο ε, περίπλοκο εξ αρχής και την περιπλοκότητά του την πληρώνουμε. Υπάρχει το τίμημα αυτής της περιπλοκότητας και θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω δράσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματι να κερδίσουμε το ποσό αυτό στο οποίο προαναφέρθηκα. Ας δώσουμε, αν μου επιτρέπετε κυρία, κυρία Πρόεδρε, το λόγο στους εμπειρογνώμονες να παρουσιάσουν τα επιμέρους θέματα στα οποία έχουν ετοιμαστεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος, για να υπενθυμίσω όλους αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν από το υπερπέραν ότι όλο αυτό το υλικό θα υπάρξει και σε εγγραφή μορφή σύντομα και φυσικά είναι και επιγραμμικά διαθέσιμο από τις διάφορες εφαρμογές για τη συνεδριάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. η πρότασή μου λοιπόν είναι να ακούσουμε τις δύο πρώτες εκθέσεις για την ελευθερία Διακίνηση αγαθών και μετά υπηρεσιών στην ενιαία αγορά και μετά να έχουμε ένα γύρο ερωτήσεων πρωτού περάσουμε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές και τις δημόσιες προμήθειες. Συμφωνείτε? Σας ευχαριστώ. Συνεχίστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την, ε, παρουσία, για την εισαγωγή και την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. παρά το γεγονό ότι η ελευθερία διακίνηση αγαθών θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα τη ενιαία αγορά, η μελέτη μα βρήκε ότι ακόμα και 20 χρόνια μετά από την θέσπιση τη ενιαία αγορά υπάρχει κατακαιρματισμό τη αγορά και ρυθμιστικά προβλήματα που εμποδίσουν την ενότητα τη αγορά. Είδαμε ιδίω να υπάρχουν προσκόμματα για, την, ε, για τις άμεσες επενδύσεις και μη δασμολογικούς φραγμούς και εμπόδια για το εμπόριο αγαθών και το δυναμικό το οποίο δεν χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους εκτιμάται σε 183-269 δισεκατομμύρια μακροχρόνια και τα αποτελέσματα αυτών των εμποδίων δεν είναι ε, ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέσαμε τρία ερευνητικά ερωτήματα στη μελέτη μας σε επίπεδο της Ευρώπης των 28. Ποια είναι τα οικονομικά ωφέλη τα οποία μπορούμε να προσποριστούμε ανάρουμε όλα τα εμπόδια στο εμπόριο στην εσωτερική αγορά. Σε εθνικό επίπεδο προσπαθήσαμε να δούμε πώς τα αποτελέσματα αυτών των εμποδίων κατανέμονται στα κράτη-μέλη. Σε τομεακό επίπεδο τέλος προσπαθήσαμε να δούμε τι θα επιτυγχάνουμε περαιτέρω εναρμόνιση σε διάφορους τομείς της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως εστιάζοντας στον τομέα των οικοδομικών υλικών. Κάποια σχόλια για αυτό το σημείο σε επίπεδο 28 μελών χρησιμοποίησαμε το οικονομικό, οικονομετρικό υπόδειγμα βαρύτητος που προσπαθεί να λάβει υπόψη τα οικονομικά ωφέλη της άρσης αυτών των εμποδίων και χρησιμοποιούμε στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, στοιχεία ΑΕΠ και στοιχεία ΩΣΑ για την ε, ρύθμιση των αγορών προϊόντων σε σχέση με τα εμπόδια αυτά και φυσικά περιλαμβάνουμε τα μη δασμολογικά εμπόδια και εμπόδια για επενδύσεις. Τι σημαίνει το υπόδειγμα βαρύτητος συνδέει το διμερές ε, εμπόριο μεταξύ δύο χωρών, στο μέγεθος της χώρας, τα εμπόδια, γεωγραφικά εμπόδια παραδείγματος χάρη όπως είναι η, απόσταση, τα πολιτιστικά εμπόδια, <clears throat> το αν έχουν μια κοινή γλώσσα ή όχι που ευνοεί το εμπόριο, στη συνέχεια τα δεσμολογικά εμπόρια και φυσικά στην εσωτερική αγορά δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο επίσης με τον ΠΟΕ έχει μειωθεί σημαντικά η σημασία αυτών των εμποδίων, αλλά σημαντικά είναι και τα εμπόδια για την ξένη άμεση επένδυση που εμποδίζουν τις εταιρείες να έχουν μετοχικό κεφάλαιο σε άλλες χώρες και να δημιουργήσουν ε, ενδιάμεσους φορείς που μπορούν να παίζουν ρόλο στα, στο εμπόριο ενδιαμέσων αγαθών και επίσης τα μη δεσμολογικά ε, εμπόδια που έχουν να κάνουν με έλλειψη αναγνώρισης, με έλλειψη εναρμόνισης και διαφορετική αντιμετώπιση φορολογία σε σχέση με ξένες εταιρείε. Σας αρέσουν οι εξισώσεις. Αυτό είναι το μοντέλο μας. Δεν θέλω να σας εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει αυτή η εξίσωση. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι βάσει αυτού του μοντέλου μη, τα μη δασμολογικά εμπόδια ε, προσκόμματα έχουν σημαντικό αποτέλεσμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιούμε τις παραμέτρους αυτής της εξίσωσης για να προβλέψουμε τι θα γίνει αν υπάρξει η άρση αυτών των προσκομμάτων για το εσωτερικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και τα αποτελέσματά μας. Υπολογίζουμε σε διάφορα σενάρια, ένα από αυτά είναι η πλήρης άρση όλων των εμποδίων και έχουμε και ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο όπου θεωρούμε ότι θα υπάρξει κάποιο επίπεδο σταθερό που βασίζεται στις πέντε χώρες που έχουν τους χαμηλότερους φραγμούς για το εμπόριο βάσει του ΩΣΑ. Εάν υπάρξει πλήρη άρση, θα ευνοηθεί το εμπόριο κατά 81 με 98 δισεκατομμύρια, 0,5% με 0,6% του ΑΕΠ. Αν αρθούν και τα εμπόδια, τα μη δασμολογικά, μπορούμε να φτάσουμε 102, 171, περίπου 0,6 έως 1% του ΑΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι αυτό είναι ένα σχετικά αισιόδοξο σενάριο, γιατί θεωρεί δεδομένο ότι όλα τα κατημέλη θα μειώσουν τους φραγμούς τους, κάτι το οποίο είναι ένα κάπως απίθανο σενάριο, αλλά σας δίνει κάποια ιδέα για το δυναμικό το οποίο δεν έχουμε ακόμα εκμεταλλευτεί για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών. Σε εθνικό επίπεδο βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα θα κατανεμηθούν ανισόμερος μεταξύ των χωρών μερών. Κάποιες από τις χώρες, οι βαλτικέ χώρες, παραγωγικά Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία θα ευνοηθούν περισσότερο από την άρση των φραγμών. Ο ΩΣΑ τονίζει ότι οι χώρες αυτές έχουν καταρχήν υψηλότερου φραγμούς για τις επενδύσει και μοιρασμολογικά εμπόδια. Σε τομεακό επίπεδο τώρα, εφαρμόσαμε αυτό το μοντέλο βαρύτητας σε επίπεδο τομεακό για τον τομέα τον κατασκευαστικό και χρησιμοποίησαμε και ένα πείραμα το οποίο έγινε ουσιαστικά όταν περάσαμε από μια οδηγία σε κανονισμό το 2013 και έχουμε τώρα πρότυπα για εναρμονισμένα προϊόντα στα κράτη-μέλη και συγκρίναμε την ε, επιρροή αυτής της αλλαγής στο εμπόριο πριν και μετά την αλλαγή σε ρυθμιστικό επίπεδο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπήρξε 3% αύξηση σε ενδοενωσιακό εμπόριο λόγω αυτής της αλλαγής σε ρυθμιστικό επίπεδο μέσα σε ένα χρόνο. Και τώρα θα ήθελα να σας παραδώσω στον επόμενο μιλτή που θα σας πει για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Ευχαριστώ.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 προκύπτει κατόπιν ε, της νομοθεσίας που υιοθετήθηκε μέσω τη Επιτροπή ΕΜΚΟ. Να το υπογραμμίσουμε και αυτό. Για τα οικοδομικά λικάνα. Ευχαριστούμε. Ε, λοιπόν, η δική μας μελέτη αφορά την ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες. Θα ήθελα αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι οι υπηρεσίες διαφέρουν πολύ από τα αγαθά Μπορούμε να γενικεύσουμε γενικά για τα αγαθά, βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά όχι στις υπηρεσίες, γιατί υπάρχει, υπάρχουν μεγάλες ε, διαφοροποιήσεις. Αυτό ήταν πάντα ένα ε, δύσκολο σημείο και για τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά και για τους νομοθέτες όπως είστε εσείς. Αρχικά λοιπόν πρέπει να θέσουμε ένα σχέδιο για την ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες, γιατί λίγοι κατανοούν πραγματικά περί τίνος πρόκειται. Μετά μιλάμε για τα κενά, θα σας τα παρουσιάσω στη συνέχεια. Λοιπόν, ο σχεδιασμός για τις υπηρεσίες. Μετά έχουμε τα έλλειμματα, σε ό,τι αφορά τον κατακαιρματισμό, αλλά έλλειμμα και ε, στην εύρυθμη λειτουργία, γιατί πολλές φορές είναι ε, έλλειμμα ανταγωνισμού και μετά έχουμε και τα οικονομικά ωφέλη. Είναι με πολύ μικρά γράμματα, δεν μπορείτε να τα δείτε από μακριά, αλλά κάποιοι από σας έχετε λάβει και έντυπο, ε, έντυπη έκδοση της μελέτης. Σελίδα 19 λοιπόν. Θα το δείτε. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται και με τους ε, CEOs της επιχειρήσης. Προσπαθούν να βάλουν ε, πολύ περίπλοκα πράγματα μέσα σε μια απλή κόλλα α4 και πρέπει να σας εξηγήσω για πάνω από ένα λεπτό ε, το πώς λειτουργεί ακριβώς η ενιαία αγορά των υπηρεσιών. Ξεκινάμε με την επικεφαλίδα της συνθήκης που περιέχει τι γενικέ υποχρεώσει από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά ελεύθερη κυκλοφορία και δικαίωμα κατάσταση, ε, πολιτική ανταγωνισμού και ευρωπαϊκά πρότυπα. Πρέπει αυτά να τα δούμε από κοινού. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο, από τα οποία προκύπτουν τα υπόλοιπα. αν αφήσουμε ένα από αυτά τα στοιχεία εκτός, ε, δεν το κατανοούμε. Μετά έχουμε το καθεστώς των οριζόντιων υπηρεσιών, το οριζόντιο μάλλον <laughs> καθεστώς υπηρεσιών, το οποίο λειτουργεί χάρη στην επικεφαλίδα ακριβώ. Αν λοιπόν ε, βασιστούμε στην οδηγία αλλά όχι στα υπόλοιπα στοιχεία, τότε δεν λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν, ε, έχουμε την οδηγία, δημόσιες προμήθειες, ε, έργα και παραχωρήσεις, υποδομές. Η εστρική αγορά πλήττεται από αυτόν τον κατακαιρματισμό της λήψης αποφάσεων και βεβαίως έχουμε και τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να πρέπει να προκύπτουν μέσω της επικορικότητας. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκού φορεί για αυτό το σκοπό που να λειτουργούν καλά. Δεν γίνεται αυτό να γίνεται στα 28 επιμέρου κρατημέλη. Γιατί αλλιώ θα έχουμε κατακαιρματισμό. Τώρα, οι επιμέρους τομεί και κλάδι το έχω διασπάσει σε έξι κομμάτια, χρηματαγορές, μεταφορές, δίκτυα, διασυνοριακές υπηρεσίε και κάποιοι ευαίσθητοι τομεί που έμειναν εκτό ε, τη οδηγία υπηρεσιών. διασυνοριακή υγεία, για παράδειγμα, έχει ε, μια ειδική οδηγία. Και τα διατομιακά καθεστώτα, ψηφιακή αγορά, λιανικό εμπόριο, όλα αυτά συνδέονται με, με ένα ευρύ φάσμα ε, διαστάσεων, γι' αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Έχουμε κάνει το δικό μας μοντέλο, γιατί η ε, έρευνα είναι ιδιαίτερα ευρεία. Λοιπόν, συλλέξαμε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. με ποσοτικά στοιχεία. Βλέπετε εδώ πέρα ότι στην οδηγία υπηρεσιών, χρηματαγορές, ε, λιανικό, ηλεκτρονικό εμπόριο και φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια έχουμε πρόσφατες και καλής ποιότητας εκτιμήσεις. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και μία έκθεση τώρα για ε, τα εμπορεύματα που μεταφέρονται για σιδηροδρόμου. Ξέρουμε ότι αυτή είναι χειρότερη, <laughs> το χειρότερο των ζωγικών είδος υπηρεσιών, αλλά πρέπει να τα δούμε όλα αυτά ε, στο γενικότερο πλαίσιο Αυτά τα εμπορεύματα λοιπόν μέσω του σιδηροδρόμου είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας και έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις ε, για τους υπόλοιπου τομείς. Κάτι θα έπρεπε να κάνουμε. Πλέον έχουμε και δεδομένα που είναι διαθέσιμα. Δυστυχώς για τις επαγγελματικές υπηρεσίες ε, είναι πολύ κακά τα στοιχεία. Δεν έχουμε καν τα στοιχειώδη δεδομένα δεν ξέρουμε πώς είναι οι επαγγελματίες ε, νομικοί που μπορούν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε στοιχεία. Και η διαδικασία της ε, συμψήφισης και της πρόσθεσης στοιχείων είναι δύσκολη. Βλέπετε εδώ τι έχουμε κάνει Έχουμε το όριο 637 δις, χαμηλότερο όριο 337, όμως από πάνω βλέπετε και μία θεά ζώνη, που, την οποία δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Είναι είτε μήπως ειδικοποιημένη, Η Επιτροπή, για παράδειγμα, σε αντίστοιχο εγχείρημα, είχε υποστοκοποιήσει τρει επιτυχίε. Ενώ πολλέ είναι σημαντικέ και υπάρχουν και άλλε που δεν μπορούμε να τι προσωπικοποιήσουμε. Δυναμικέ επιπτώσει που όμω ε, μα επηρεάζουν. Πολύ πάνω λοιπόν από τα 67 πάμε, αλλά δεν μπορώ να σα πω πόσο. Και τέλο. Εδώ πέρα επειδή μπερδεύουμε διαφορετικά πράγματα, πρέπει να λάβουμε πολλά πράγματα υπόψη. Κατανοώ ότι οι Ευρωβουλευτές θέλουν να ακούσουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Να θέσετε ερωτήματα και θέλετε να ακούσετε όλες τις ε, παρουσιάσεις πρώτα. Ας συνεχίσουμε. Εντάξει. Τώρα ερχόμαστε στις δημόσιες προμήθειες. Μάλλον στην ψηφιακή η αγορά. Uh, uh, uh, Σας ευχαριστώ. Θα αναφερθώ στην μελέτη για την ψηφιακή αγορά και ιδιότερα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η προσέγγιση μας είναι ότι προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η νομοθεσία που θεσπίζει την ψηφιακή αγορά, να δούμε πού υπάρχουν δυνητικά κενά και ελλείψεις, να δούμε πώς εφαρμόζεται στην πράξη, ποια είναι τα κενά στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και βλέπουμε το, προσπαθούμε να δούμε πόσο, πώς μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε το κόστος το οποίο συνοδεύει αυτή την νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά τα κενά, υπάρχουν τρεις τομείς όπου μπορούμε να έχουμε σχετικά λογικούς, ε, λογικές ε, εκτιμήσεις. Καταρχήν το υπολογιστικό νέφος γιατί δεν υπάρχει ε, η αστική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Όταν λέτε βάλτε τα δεδομένα σας εκεί, δεν είναι καθόλου σαφές ποιος είναι ο υπεύθυνος για την ακαιρεότητα των δεδομένων και την προστασία τους. Υπάρχει ο τομέας των πληρωμών, των ηλεκτρονικών πληρωμών, όπου δεν υπάρχει μεγάλο χάσμα στις νομοθεσίες αλλά υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές σε εμπορικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών. Λόγω των διαφορετικών συστημάτων χρηματοοικονομικών που ίσιαν στα κράτη-μέλη. Και όλα αυτά κάνουν τις διαμεθοριακές πληρωμές πιο πολυδάπανες από ό,τι για τις εσωτερικές πληρωμές. Ένας τρίτος τομέας που εξετάζουμε είναι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες γραμμάτων και δεμάτων. Πολλά λοιπόν αγαθά μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο, παραδίδονται στους ε, τελικούς αγοραστές με τον τρόπο αυτό. Και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα με έλλειψη νομοθεσίας, αλλά το πρόβλημα οφείλεται στην έλλειψη πληροφοριών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα ορισμένων ε, επιλογών και με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο πολυδάπανη η παράδοση με το ταχυδρομείο και δημιουργούνται εμπόδια για τη μεθοδιακή διαμεθοριακή λειτουργία των ταχυδρομείων. Άλλα δυνητικά κενά, ίσως πιο σημαντικά, τα οποία δεν τα αντιμετωπίσαμε ποσοτικά. Ένα παράδειγμα, η ηλεκτρονική υπογραφή. Είναι ένας τομέας όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί περισσότερο περιθώριο για αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Θα μπορούσαν να υπάρξουν σημαντικά κέρδη λοιπόν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής. Αλλά δεν είναι εύκολο εδώ να κάνουμε ένα λογικό υπολογισμό, μια λογική εκτίμηση του κέρδους που θα μπορούσε να προκύψει. Για να πάτε μια ιδέα για τα ποσοτικά μεγέθη, μιλάμε για 50 με 60 δισεκατομμύρια και το μεγαλύτερο μέρος έχει να κάνει με το υπολογιστικό νέφος. Έχουμε ένα δεύτερο επίπεδο όπου προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εκτιμήσεις κόστους και να τις ενσωματώσουμε σε ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε τι μπορεί να επιτευχθεί με το κλείσιμο αυτών των χασμάτων. Τα αποτελέσματά μας ε, δίνουν την εντύπωση ότι θα μπορούσε να κερδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 0,4% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 και θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και περίπου 220.000 θέσεις απασχόλησης. <clears throat> Βέβαια αυτό είναι μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω και τα στοιχεία αυτά μονάχα ε, αφορούν τα χάσματα στους τρεις αυτούς τομείς όπου έχουμε κάποια δυνατότητα ποσοτικοποίησης. Δεν είναι το συνολικό κέρδος το οποίο θα μπορούσε να προκύψει από την εναρμόνιση. Τα συμπεράσματά μας είναι Φυσικά <clears throat> ενισχύεται η ψηφιακή αγορά και όλο και περισσότερο διασυνδέεται με την παραδοσιακή οικονομία. Επομένως όλο και περισσότερο θα είναι σημαντική η ψηφιακή οικονομία. Δεύτερον, υπήρξε σημαντική νομοθετική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια που κάνει πιο δύσκολη βέβαια για την αξιολόγηση της κατάστασης και θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ευφυής παρακολούθηση για να μπορέσουμε <clears throat> να εντοπίσουμε το, το κατά πόσο η νομοθεσία αυτή αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία την προκάλεσαν. Μια άλλη παρατήρηση, ίσως σε πολλούς από αυτούς τους τομείς υπάρχουν και μη νομοθετικού χαρακτήρα ρυθμίσεις οι οποίες μπορεί να είναι ελπιδοφόρες εθελοντικές συμφωνίες και δεσμεύσεις για πρότυπα. Μπορεί να βοηθήσει λοιπόν κάτι τέτοιο γιατί αναπτύσσεται τόσο γρήγορα αυτό ο τομέα που υπολείπεται πάντα η νομοθετική ρύθμιση πίσω από την τεχνολογική ανάπτυξη. Και προφανώς βέβαια τα στοιχεία λοιπόν αυτά που έχουμε εκτιμήσει αφορούν τρεις τομείς μονάχα, αλλά σίγουρα μιλάμε για σημαντικό οικονομικό κόστος. Ευχαριστώ. And were you also giving the presentation on consumers and public procurement? Μπορείτε να μας κάνετε την παρουσίαση για τους καταναλωτές και τις δημόσιες προμήθειες. Okay, good morning. Um, I'm going to speak to you today about the cost of non-Europe in the case of public... Λοιπόν, ο κόστος της μη Ευρώπης στον τομέα των δημοσίων προμήθειων. Να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι παρουσιάστηκαν οι γενικότεροι στόχοι της έρευνας, το κόστος των κενών στην νομοθεσία στον τομέα των δημοσίων προμηθειών και εκχωρήσεων και ανάλυση των ωφελημάτων από την κοινή αγορά. Τέσσερα στοιχεία λάβαμε υπόψη μας. Πρώτον, εξετάσαμε το τι πηγές γραπτές έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα σχετικά με τον υπολογισμό του κόστους και του οφέλους και κάναμε μία επιλογή αντιπροσωπευτικών μελετών κατά περίπτωση, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε στην μελέτη μας. Δεύτερο στοιχείο ήταν η έρευνα την οποία κάναμε επιγραφείου σε εισαγωγικά, Προσπαθήσαμε δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας σε επίπεδο οικονομικών αναλύσεων, εγκάρσιων μελετών, οριζόντιων μελετών. Ε, τρεις περιπτώσεις επιμέρους μελετήσαμε, οι οποίες νομίζω αντικατοπτρίζουν σωστά τα προβλήματα τα οποία έχει η ε, νομοθετική ρύθμιση ισχύουσα στον τομέα των δημοσίων ε, διαγωνισμών, προμηθειών κτλ. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς αλλά και η δημόσια διοίκηση που θέτει σε λειτουργία αυτές τις διαδικασίες. Και τέλος κάνουμε μια οικονομική ανάλυση προσπαθώντας να ποσοστικοποιήσουμε τα ωφέλη αλλά και το κόστος των ε, κενών που διαπιστώνονται σήμερα. Καταρχάς τα κενά τα οποία εντοπίσαμε στον τομέα που μας ενδιαφέρει. Πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για κενά τα οποία ίσχυαν πριν από τη νέα νομοθεσία η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Μας ζητήθηκε μια evidence-based study. Προσπαθήσαμε δηλαδή να συλλέξουμε επιμέρους στοιχεία και τεκμήρια. Κάναμε λοιπόν μια ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας, των στόχων που θέλουμε να πετύχουμε και όλα αυτά βασίζονται βέβαια σε κενά που υπήρχαν πριν από την εισαγωγή της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης στην αρχή ε, του ε, χρόνου. Έξι τομείς εντοπίστηκαν στους οποίους ε, πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις, η εμβέλεια της οδηγίας, οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται, κάποιες επιλογές που είναι στη διάθεσή τους και όχι μια γενική ισχύω διαδικασία, Υπήρξαν κάποιες ανησυχίες για την απαιτούμενη και επιθυμητή ευελιξία σε επίπεδο διαδικασιών, κάτι το οποίο αντιμετωπίζει η νέα νομοθεσία. Τώρα για στρατηγικής φύσεως προμήθειες, εδώ συμπεριλαμβάνουμε και τους περιβαλλοντικούς στόχους και υπάρχουν κίνδυνοι σε σχέση με αυτό και σε σχέση με αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σε τομείς οι οποίοι στο παρελθόν τουλάχιστον ετύχαναν διαφορετικής μεταχείρισης. Τώρα πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες, εδώ τίθεται το θέμα των γλωσσών που χρησιμοποιούνται, οι συνεννοήσεις ανάμεσα σε δύο μέρη, σε διαφορετικές χώρες και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών σε επίπεδο νομοθετικό. Όλα αυτά λοιπόν ίσχυαν μέχρι τις αρχές του χρόνου και εν μέρη έχουν αντιμετωπιστεί. Οι παραχωρήσεις τώρα σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς περισσότερο έχουν κάποια σημασία. Λοιπόν, εδώ είναι τα ευρήματά μας, κάποια από αυτά σε σχέση με το διοικητικό κόστος, με την έλλειψη κατανόησης που πολλές φορές έχουμε για τις ακολουθητές διαδικασίες και για την αβέβαιη χρήση από πλευράς των αρχών των κανόνων. Αντιμετωπίσαμε δύο τρόπους ποσοτικής ανάλυσης. Ο πρώτος ε, τρόπος βασίστηκε στη μελέτη που ξεκίνησε το 2006 και βρήκαμε ακριβώς ποια ήταν τα ωφέλη τότε. Χρησιμοποιώντας αυτές τις ε, εκτιμήσεις έχει από τότε μεγαλώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν μεγαλώσει και οι δαπάνες στον τομέα των δημοσίων δαπανών και δημοσίων μάλλον διαγωνισμών και προμηθειών Είχαμε δει ποιο ήταν η αρχική διαπίστωση τσεκίνη και το κενό τσεκίνη όπως λέγαμε τώρα και είχαμε πει ότι το κόστος της μη Ευρώπης είναι γύρω στα 50 δις. Έχουν όμως υπάρξει εκτιμήσεις εξιολόγησης, εξοικονόμησης συγγνώμη, ποσών πιστώσεων που φτάνουν τα 23 περίπου δις. Νομίζω ότι και στις τρεις περιπτώσεις τις οποίες μελετήσαμε προσπαθήσαμε εγκάρσια να εξετάσουμε τις επιπτώσεις και φτάσαμε περίπου ε, εκ των κάτω προς τα πάνω σε ένα υπολογισμό περίπου 57,3 δις. Λοιπόν, στα συμπεράσματά μας εμείς βασιζόμαστε στην γενική εκτίμηση την οποία κάναμε ότι υπάρχει μια εξοικονόμηση πιστώσεων 22,7 δις. Κάποια από τα κενά τα οποία υπήρχαν πριν από το 2014 θα καλυφθούν από τη νέα νομοθετική ρύθμιση εν μέρη. Δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακόμα αυτό, αν και αυτό πιστεύουμε ότι σε έφθετο χρόνο θα γίνει πραγματικότητα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά τα οποία δεν θα καλυφθούν όλα. Είναι φυσικά εμπόδια τα θέματα τα γλωσσικά σαν παράδειγμα, είναι σαν φυσικά εμπόδια. Υπάρχουν επίσης κάποιες υπηρεσίες ε, οι οποίες ε, είναι πολύ λογικότερο να παρέχονται τοπικά. Εν πάση περιπτώσει εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης και σίγουρα οι τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις σαφώς θα βελτιώσουν την κατάσταση. Thank you, Ευχαριστούμε, Chris. Να δώσουμε και πάρα το λόγο στο Βόιτσεκ για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ πολύ. Ένα συνάδελφο την έκανε πραγματικά τη μελέτη, αλλά δεν κατάφερε να παρευρεθεί σήμερα, οπότε τον αντικαθιστώ. Η προσέγγιση είναι παρόμοια. Προσπαθούμε να εξετάσουμε την νομοθεσία στον τομέα του ε, και ακτιμένου των καταναλωτών και θέλουμε να εντοπίσουμε πιθανά κενά στην ομοθέσια, αλλά να βρούμε και πρακτικούς ε, τρόπους ε, με τους οποίους ε, επηρεάζονται καταναλωτές και επιχειρήσεις από αυτά τα κενά. Και πάλι βάσει αποδεικτών στοιχείων και δεδομένων θέλουμε να βασιστούμε σε αυτά λοιπόν για να διαμορφώσουμε μία νέα προσέγγιση. Ποια είναι αυτά τα κενά λοιπόν στον τομέα του καταναλωτικού κεκτημένου, σε αρκετού τομεί θεωρούμε ότι μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοια. Για παράδειγμα, εμπορικές εγγύησει, όταν έχουμε κατακαιρματισμό σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη εφιστάμενη νομοθεσία. Κάποιοι άλλοι τομείς δεν καλύπτονται από την νομοθεσία. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε συναλλαγέ όπου ο καταναλωτή, ε, πολλοί αντικείμενα σε έμπορο, όπως για παράδειγμα αντίκες, αντικείμενα υψηλής αξίας, αλλά σε σκιώτες αγορές. Μετά έχουμε συναλλαγές από καταναλωτή σε καταναλωτή, χωρίς ε, διαμεσολαβητή ή μεσάζοντα. Ε, συνήθως ε, αυτό αφορά ε, επιγραμμικά μέσα όπως είναι το eBay. Μετά έχουμε τον ε, τομέα των καταναλωτικών δανείων όπου η προστασία είναι άνηση και πολλές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου δεν είναι υποχρεωτικές. Και μετά έχουμε και τον τομέα ε, των ε, τυχερών παιχνίων και στο διαδίκτυο, όπου υπάρχει έλλειψη προστασίας από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτά είναι τα κενά που προσπαθήσαμε να ποσοτοκοποιήσουμε και πιο συγκεκριμένα εστιαστήκαμε σε τρεις εμπορικά εχέγγυα, καταναλωτικά δάνεια και τυχερά παίγνια στο δίκτυο και εκτός. Και τα στοιχεία στα οποία καταλήξαμε είναι τα υψηλότερα στον τομέα των παιχνίων. Το συνολικό κόστος είναι περίπου 5,5 δις ευρώ και συνδέεται κυρίως με τις ε, πολύμορφες ε, προϋποθέσεις που θέτουν ε, οι αρχές των επιμέρους κρατών μελών. Επομένω, η θέσπιση μιας ενιαίας αγοράς θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε σύγκληση σε αυτόν τον κλάδο. Και η δεύτερη πτυχή αφορά τους εθισμένους στα τυχερά παίγνια. Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση μέσω της ε, επίτευξης της ενίας αγοράς. Για τα καταναλωτικά δάνεια είναι χαμηλότερα τα στοιχεία, κυρίως επειδή έχουμε περισσότερο δυσυνοριακό ανταγωνισμό, κάτι το οποίο οδηγεί και πάλι στη σύγκληση των ε, καταναλωτικών όρων. ένα ξεχωριστό εγχείρημα ήταν να υπολογίσουμε ποιο θα ήταν το πιθανό ε, όφελος αν κλείσουμε όλα αυτά τα κενά και καταλήγουμε ε, στο ποσό των 58 δις ευρώ. Συμπερασματικά και πάλι το κατανοητικό κεκτημένο ε, είναι ένα μέσο που έχει υπάρξει σημαντική νομοθετική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Έχει αυξηθεί η προστασία των ε, ε, καταναλωτών και η ισχύ του. Παραμένουν βέβαια κάποια νομοθετικά κενά και θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη δραστηριότητα νομοθετική, ιδίω εκεί όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά όπω είναι ο τομέα των ε, τυχερών παιχνίων. Κατανοούμε βεβαίω ότι είναι και κάποια δύσκολα στοιχεία εδώ. Μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι ε, είναι, υπάρχει πολύ στενή σύνδεση και με άλλους ε, νομοθετικούς τομείς. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε και την ευρύτερη εικόνα για το πώς το καταναλωτικό κεκτημένο θα ε, επηρεάσει την προσέγγιση μας, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ε, ψηφιακή έννοια αγορά, τις υπηρεσίες και το καθεξής. Και τέλος, η τεχνολογία και τα ε, μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά μοντέλα πολύ συχνά υποχρεώνουν την νομοθεσία να τους προλάβει εκ των υστέρων. Ευχαριστώ πολύ. I, Ίσως θα πρέπει να το έχω κάνει αυτό στην αρχή και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν ήμουν σαφής για το ποιος κάνει την, ποια παρουσίαση για να ξέρετε σε ποιον θα απευθύνεται τα ερωτήματα το κόστος της μη Ευρώπης για τα αγαθά ο Μάρκος Χάφνερ επί υπηρεσίες ο Ζακ Πέλκμανς από το ΣΕΠΣ Ο Κρίς Σμιθ έκανε την παρουσίαση για τις δημόσιες προμήθειες από τη Europe Economics και ακούσατε τον Βόιτσεκ Πεζίνσκι, αν το προφέρω σωστά, από την GHK International που αναφέρθηκε στην ψηφιακή ενιαία αγορά και για το κεκτημένο σε επίπεδο καταναλωτών. Έχετε τώρα στους φακέλους σας την πλήρη ε, παρουσίαση αυτών των μελετών. Κάποιες από αυτές, θα, κάποια κομμάτια τους θα μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες, αλλά αυτό μοναχά αν το ζητήσετε, γιατί αυτό ήταν κάτι που ζήτησε η Επιτροπή μας. Είναι δικές μας εκθέσεις. Θα ήθελα να σας ζητήσω να τις αναδυφίσετε γιατί οι παρουσιάσεις που ακούσατε σήμερα ήταν υψηλού επίπεδου και οι μελέτες αυτές έχουν πολύ λεπτομέρεια. και ίσως είναι κάπως ε, παραπλανητικά τα στοιχεία γιατί οι παρουσιάσεις για τις, ε, την ψηφιακή Ευρώπη και τις, δημόσιες, και τις προμήθειες είναι στο ίδιο σημείο στο φακελό σας αλλά οι επιμέρους μελέτες για τις υπηρεσίες που αναφέρατε έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τον ιωτικό εξοπλισμό που τονίζει και τη σημασία του να είναι προσβάσιμα οικονομικά τα προϊόντα αυτά και υψηλής ποιότητος και να είναι εύκολα <clears throat> διαθέσιμα. Δεν είναι μοναχά θέμα λοιπόν κόστους, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και απασχολεί πολλούς από τους πολίτες μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη που ξεκινάει στη σελίδα 53 για την ε, μελέτη για την ενιαία αγορά και τα άγαθα. Μπορείτε λοιπόν να δείτε λεπτομεριακά μερικές από αυτές τις μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων που είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Ε, Μαρία Κουκίν θέλω να θέσει ένα ερώτημα τώρα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. πολύ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που θέσατε το θέμα αυτό προς συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους εμπειρογνώμονες που παρουσίασαν κάποιες εκθέσεις πολύτιμες για, τις εσωτερικές αγορά, για την εσωτερική αγορά. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για αυτούς να παρουσιάσουν όλη τους την εργασία μέσα σε λίγα λεπτά. Θα τα διαβάσω πολύ προσεκτικά για τη δική μου χώρα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δυστυχώς δεν έχω τα ονόματά σας σωστά, αλλά νομίζω θα καταλάβετε σε ποιους απευθύνεται κάθε φορά η ερώτησή μου. Πρώτον, η ενιαία αγορά αυτή τη στιγμή φύγεται από πάρα πολλά αρνητικά χαρακτηριστικά. Δεν αναφερθήκατε πάρα πολύ για το εξής θέμα. Οι αποδείξεις πληρωμών που είναι διαφορετικές από τη μία χώρα στην άλλη και δημιουργούν σύγχυση. Ε, πώς θα αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο. Αυτά οι αποδείξεις πληρωμών όταν έρχονται στην αγορά δεν γίνονται άμεσα αποδεκτές μερικές φορές. Αναφέρομαι στις αποδείξεις όπως είπα για την πληρωμή μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Μια επιπλέον ερώτηση. Στις μελέτες σας έχετε αναλύσει επίσης τις ε, συμβάσεις αγοραπολισιών που διατυπώνονται με διαφορετικό τρόπο αναχώρα ένα παράδειγμα, αν έχουμε έναν Ρουμάνο παραγωγό ο οποίος θέλει ε, να πωλήσει κάτι μέσω της αλυσίδας καταστημάτων μετρό. Θα πρέπει να υπογράψει μία σύμβαση στη Ρουμανία, μία σύμβαση στη Γερμανία, μία σύμβαση σε τρίτη χώρα. Το διοικητικό κόστος και το κόστος διαχείρισης αυτών των συμβολέων, των συμβάσεων μάλλον, είναι ιδιαίτερο υψηλό. Ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειες. Η χώρα μου εδώ χαρακτηρίζεται από τεράστιες καθυστερήσεις και οι δυνατότητες αμφισβήτησης του αποτελέσματος μιας διαδικασίας επιλογής είναι πολύ περίπλοκοι και μακροπρόθεσμοι. Λοιπόν, αυτές τις καθυστερήσεις 6 ενός έτους και περισσότερο ε, είναι κάτι το πάρα πολύ ε, προβληματικό γιατί πολλές φορές οι αφισβητήσεις έχουν κακή πρόθεση. Είναι ένα είδος διαφθοράς και αυτό. Δεν ακούω. Η κυρία Γιάκον Σάρη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η αριθμή αυτή πράγματι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες. Αν πράγματι απλουστεύσουμε τα πράγματα και αν μπορέσουμε να καταστήσουμε λειτουργική την εσωτερική αγορά, νομίζω ότι ταυτόχρονα θα έχουμε βρει την λύση για την κρίση. Εάν βάλουμε την προτεραιότητα στα θετικά, αν ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας ρωτήσει ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα στα οποία πρέπει να παρέμβουμε για να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά, τι θα πείτε. Ποια θα είναι η απάντησή σας. Και πώς μπορούμε να συνδέσουμε την διόρθωση όλων αυτών των κενών και τις προτεραιότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει για κάτι άλλο το οποίο μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον σε επίπεδο περιφερειακό. Βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε διάφορες χώρες ή και μέσα σε χώρες όπως η Ισπανία είναι μια χώρα αν καλά ε, θα ωφεληθεί λιγότερο. Για ποιο λόγο δεν το καταλαβαίνω. Ε, Παρ' όλα αυτά έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα σας και τέτοιες ερωτήσεις όπως αυτές που θέτω τώρα τίθενται. πολύ συχνά μας λέγουν ε, γιατί ε, έχουμε λόγο να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα μας δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορούμε να απαντούμε σε τέτοιες ερωτήσεις. Μια τρίτη ερώτηση και μετά θα δώσετε απάντηση και στις τρεις από κοινού. Και μετά ε, μια δεύτερη και μια τρίτη. Κοέλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω αυτούς που έχουν κάνει τη μελέτη αυτή, που συνεχίζει το έργο του καθηγητού Τσεκίνη και που αντιμετωπίζει ένα σύνολο πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα μπορέσει να μας βοηθήσει να ανοίξουμε καινοτόμους δρόμους στην Ευρώπη ακολουθώντας τη λογική της έκθεσης εκείνης στο παρελθόν. Είναι γεγονός ότι όλες οι χώρες δεν θα έχουν το ίδιο όφελος. Αυτό μας αναγκάζει να αναλύσουμε και πολιτικά πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ισοδίκαια μεταχείριση όλων των χωρών, αλλά είναι γεγονός ότι όλες οι χώρες μπορούν να κερδίσουν κάτι με την υπέρβαση των φραγμών. Γιατί αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ είναι η άρση των φραγμών αυτών, ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλοι καλύτερα την εσωτερική αγορά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ε, τους εξής λόγους. Πρώτον, ότι είμαστε, όπως είπαν οι συνάδελφοι, σε μια φάση κρίσης και οτιδήποτε δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης θα πρέπει να το προωθήσουμε. Και δεύτερον, έχει ένα πολιτικό χαρακτήρα το θέμα αυτό. Όταν λένε ορισμένοι ότι χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη για πιο εθνική αντιμετώπιση, αυτή η μελέτη καταδεικνύει ακριβώς το αντίθετο, ότι χρειαζόμαστε πράγματι περισσότερη Ευρώπη, τουλάχιστον στον τομέα αυτό και πρέπει να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια που εμποδίζουν την Ένωση στο οικονομικό επίπεδο. Ήθελα τώρα να έρθω στο σημείο των καταναλωτών. Εκεί εκτιμάται ότι θα μπορεί να υπάρξει μεγάλη βελτίωση και μεγάλο κέρδος σε ό,τι αφορά τον επιγραμμικό τζόγο, τα τυχηρά παιχνίδια. Και εδώ δεν βλέπω μία σύνδεση μεταξύ αυτών που λέγονται στην έκθεση, τα διάφορα τμήματα του κέρδους που αναφέρονται και το τελικό συμπέρασμα. Υπάρχουν ορισμένοι αριθμοί και υπάρχει το προστοκόμενο όφελος των 58 δισεκατομμυρίων. Πώς έφτασαν οι συντάκτες έκθεση σε αυτό το τελικό ποσό τη στιγμή που από τα διάφορα τμήματα δεν φαίνεται να φτάνουμε σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα των τυχερών παιχνιδίων. Can we take those first three? Να απαντήσουμε σε αυτές τις τρεις πρώτες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να δώσω κάποιες πρώτες απαντήσεις εγώ και μετά αν συμφωνείτε μπορούν να προσθέσουν και την άποψή τους και οι εμπειρογνώμονες. Για να απαντήσω στην κυρία Γκραπίνη επιγραμματικά σε ό,τι φορά τα τιμολόγια τα, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αν κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ε, θα έχουμε τεράστια οικονομικά ωφέλη. Οι εμπειρογνώμονες μπορούν να σας δέσουν περισσότερα στοιχεία. Για τις ε, συμβάσεις ε, πωλήσεων, αυτό είναι θέμα ιδιωτικού διεθνού δικαίου και για τις καθυστερήσεις στις δημόσιες προμήθειες. Να σας παραπέμψω στην νομοθεσία περί καθυστερημένων πληρωμών που πέρασε από την ΙΜΚΟ Είχαμε και μία ε, διάσκεψη υπό την Ιταλική Προεδρία για αυτό το θέμα και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για αυτή την Επιτροπή να εξετάσει πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία. Γιατί όταν υιοθετήθηκε η νομοθεσία, όπως είπε η κυρία Γκραπίνη, ήταν σαφές ότι ε, υπήρχαν τεράστιες απώλειες επιχειρήσεις ε, κήρυσαν πτώχευση ακριβώς λόγω των καθυστερήσεων. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υιοθετήθηκε αυτή η νομοθετική πράξη αλλά από ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά τα πράγματα. Θα ήταν λοιπόν μια καλή ευκαιρία η Επιτροπή σας ε, να κάνει κάτι γι' αυτό και εμείς βεβαίως ε, να βοηθήσουμε. Για την κυρία Γιακονσάρη, να πω ότι και μένα τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία θα είναι η ενιαία ψηφιακή αγορά και η αντιμετώπιση του φαινομένου του ε, ε, ρυθμιστικού κατακαιρματισμού. Αυτό συνδέεται και με τις ευφυείς ρυθμίσεις, το καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο και το καθεξής. Γιατί έτσι βεβαίω πάντα μπορούν να ανακύψουν νέα εμπόδια, όμως θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την καλύτερη ροή της αγοράς. Ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, ξεπερνούνται προβλήματα μέσω ε, συμφωνιών σε εθελοντική βάση. Πρόσφατες μελέτες, όπως από Μορέτη και Κοριτσέλη, φέτος μάλιστα, δείχνουν ότι, για να απαντήσω στον κύριο Κοέλιο, όλα τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κέρδισαν τουλάχιστον 10% ε, στο ΑΕΠ τους. Και μάλιστα αυτό ε, το αποτέλεσμα αυξάνεται συνεχώς. Η μοναδική εξαίρεση είναι η Ελλάδα. Γιατί το ΑΕΠ δεν έχει αυξηθεί με τον ίδιο τρόπο μετά από την ένταξή της. Μπορούν οι περιογνώμονες ε, να αναφερθούν περαιτέρω, αλλά νομίζω ότι δεν το έχουμε μελετήσει αρκετά. Θα πρέπει να το εξετάσουμε και για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο δεν προτείνουμε να υπάρχει νομοθεσία. Ξέρω πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το ζήτημα. Απλώς η ενιαία αγορά στα τυχερά παιχνίδια θα έχει οικονομικά ωφέλη. Μπορεί να εξηγήσει παραπάνω ο εμπειρογνώμονας. Αυτά από μένα. Πρόεδρε. Να πω μόνο ότι έχουμε ακόμα 8 ερωτήσεις. Επομένω, αν μπορείτε να απαντήσετε εν συντομία. Το βασικό ζήτημα που θα μπορούσα τουλάχιστον να προσπαθήσω να απαντήσω είναι ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες. Τι να πούμε στο Γιούγκερ. Πρέπει να βρούμε ποια είναι η κύρια δυσκολία. Γιατί είναι το γνωστό θέμα με το ελαττήριο. Όσο, πιο, όσο το σπρώνεις προς τα κάτω, τόσο πιο δύσκολο είναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλέ ατέλειε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ή δεν μπορούμε να αποστοκοποιήσουμε. Όπω και να έχει όμω, αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι πολύ ψηλά. Ακόμα και έξω να έχουμε πέσει και να είναι πολύ χαμηλότερα, πάλι θα είναι πολύ ψηλά. Έχουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο του ελατηρίου. Και γιατί ισχύει αυτό. Πρώτον, οδηγία περιπηρεσιών. Αν ήσασταν εδώ πριν 7-8 χρόνια, στην Επιτροπή Ημικό εδώ, τα καταλαβαίνατε. Ένα από τα πολύ καλά στοιχεία κατά τη γνώμη μου, ή μάλλον αυτό που προκαλούν έκπληξη, είναι ότι υπάρχει σιγή ηχθείως για αυτή την οδηγία. Είναι επιτυχία η οδηγία υπηρεσιών, ναι. Αρκεί, μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω πράγματα από, από, με αυτό, ναι, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες, όπως είναι επαγγελματίε, για αυτη την οδηγια ειναι επιτυχια η οδηγια υπηρεσιων ναι αρκει μπορουμε να κανουμε και παραπανω πραγματα απο με αυτο ναι αλλα υπαρχουν και δυσκολιες οπως ειναι επαγγελματιε για παραδειγμα Δεύτερον, βιομηχανίες δικτύων. Μπορεί να μην αφορά την Επιτροπή σας, αλλά εμείς το εξετάζουμε συνολικά. Για την αγορά ενέργειας, η πίεση είναι πολύ πιο μεγάλη όταν πιέζει ο κύριος Πούτιν παρά όταν πιέζουν οι ευρωπαϊκές αρχές ή οποιοδήποτε άλλος. Ας είμαστε ειλικρινείς εδώ. ηλεκτρονικό εμπόριο και σιδηροδρομικά δίκτυα είναι υπηρεσίες δικτύων. Και εκεί δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ε, διατάξεις, είτε δεν τις θέλουμε. Κάτι άλλο το οποίο αφορά τα δίκτυα είναι οι υποδομές. Αυτά δεν έρχονται έτσι από μόνα τους. Αν θέλουμε πραγματική ενιαία αγορά στην ενέργεια ε, και στις υποδομές και στο σιδηρόδρομο θα πρέπει να επενδύσουμε. Πολύ μαζικές επενδύσεις ε, στο σιδηρόδρομο αλλά και γενικά. Μετά, ιδιωτικό δίκαιο επισήμως είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δημιουργεί και προβλήματα μετά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι ε, πωλήσει, καταναλωτικά ζητήματα, παρότι έχει σημειωθεί ο πρόοδο, εδώ παραμένει το θέμα, και ψηφιακή ενιαία αγορά. Αν δείτε τα 137 σημεία στον κατάλογο τη κυρία Κλού, τα μισά, αν όχι παραπάνω, αφορούν ζητήματα ιδιωτικού δικαίου. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο. Μπορούμε να το κάνουμε, ναι. Αλλά μετά υπάρχει και η ε, ρυθμιστική ετερογένεια συχνά προκαλείται από τα κράτη-μέλη που κάποιες φορές παράτυπα περνούν τη δική τους νομοθεσία. Δεν τα λέω όλα αυτά για να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά για να τα γνωρίζουμε καλύτερα. Βέβαια θα είναι πολύ καλό να καταφέρουμε να πιέσουμε το τελατήριο προς τα κάτω, αλλά χρειαζόμαστε εμεί για να το κάνουμε αυτό. Θα ήθελα να απαντήσω για ένα συγκεκριμένο σημείο υπήρχε ένα ερώτημα για τα στοιχεία σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Υπάρχει μια διαφορά σε προσέγγιση. τα τυχερά παιχνίδια ήταν μία από τις επιμέρους περιπτώσεις που ερευνήθηκαν ενώ το συνολικό ποσό είναι μία άσκηση εκ των άνω προς τα κάτω προσπαθούμε να δούμε το σύνολο για τους καταλαβητές. Επομένως οι δύο προσεγγίσεις αυτές δεν είναι εύκολα συνδυάσιμες. το όφελος το οποίο έχει εντοπιστεί βασίζεται κυρίως στην ε, σύγκληση των ε, ρυθμίσεων σε σχέση με τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, γιατί ξέρετε ότι δουλεύουν διαφορετικά αυτά στα διάφορα κράτη. Και επίσης το θέμα της μείωσης του κόστους που προέρχεται από τους προβληματικούς ε, τζογαδόρους. Είναι πολύπλοκα λοιπόν όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να τα εξηγήσει κανείς. Αν θέλει κανείς πάντως να σκεφτεί για νομοθετική δράση στον τομέα αυτό, θα χρειαζόταν περισσότερο σε βάθος ε, μελέτη. Εγώ θα απαντήσω εν συντομία σε ορισμένε ε, ε, προτάσεις που έγιναν σε σχέση με την διακίνηση αγαθών. Εμείς έχουμε κάνει ποσοτική εργασία στη μελέτη μας, αλλά προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και πιο ποιοτικά και ήρθαμε σε επαφή και κάναμε συνεντεύξεις με πολλούς ε, καταναλωτές, με μικρομεσαίες επιχείρησεις, να δούμε ποια είναι τα προσκόμματα στην ενιαία αγορά αγαθών. Αυτό το οποίο είδαμε ότι πράγματι πλήττονται από την καθυστέρηση ή τη μην έγκριση εναρμονισμένων κανόνα για τα αγαθά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν έχουν πολλαπλά πρότυπα με τα οποία πρέπει να συμμορφωθούν, αυτό είναι σχετικά πολύ δάπανα αν θέλουν να λειτουργήσουν σε πολλές αγορές. <clears throat> Μια ενδιαφέρουσα πτυχή εδώ είναι η, αν θέλετε, το πλεονέκτημα έδρας, ότι ο καταναλωτής προτιμάει να αγοράζει τα προϊόντα από τη χώρα του, από ότι από άλλες χώρες και αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα για το διενοσιακό εμπόριο. Μία επιλογή που είδαμε για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα είναι να ευνοήσουμε <clears throat> το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων κυρίως και μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων με σαφείς κανόνες οι οποίοι σιγά σιγά θα καλύψουν τα κενά της ενιαίας αγοράς. Αυτά λοιπόν εν συντομία για το πού μπορούν να υπάρχουν επιλογές σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, αλλά δεν έχουμε βρει μια πανάκια, ένα ενιαίο τρόπο για να ξεπεράσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα όλα αυτά τα εμπόδια. Για τις περιφερειακές διαφορές. Η μελέτη μας βασίστηκε σε στοιχεία του ΟΣΑ και τα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να προκύψει κέρδος για όλες τις χώρες αν υπάρξει άρση των εμποδίων στο εμπόριο. Για κάποιες χώρες που είχαν αρχικά υψηλά εμπόδια θα μπορέσουν να συγκλίνουν με τον τρόπο αυτό και θα κερδίσουν φυσικά περισσότερο σε πρώτο στάδιο από την άρση αυτών των ε, προσκομμάτων. Νομίζω ότι έτσι μπορώ να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που τέθηκαν. Λάγκεν, Στέφανης Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήταν εξόχως ενδιαφέρουσες αυτές οι εκθέσεις και κατέληξαν πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και ιδίως της ψηφιακής αγοράς. Με εντυπωσιάζει πόσες ευκαιρίες παραμένουν ακόμα και πόσα εμπόδια παραμένουν ακόμα στην ψηφιακή αγορά. Εκεί λοιπόν πρέπει να τεθεί η έμφαση τα επόμενα χρόνια αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη και απασχόληση για την Ευρώπη, που είναι ο στόχος όλων μας. Ένα μικρό ερώτημα. Είπατε ότι από τις πέντε διαφορετικούς αυτούς τομείς μπορεί να προκύψει 5 8% αύξηση του ΑΕΠ. Το ερώτημα είναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σωρευτικό και υπάρχουν πραγματικά συνέργειες μεταξύ των τομέων αυτών που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τους εντυπωσιακούς αριθμούς που μας δώσατε, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών. Βασική μου ερώτηση είναι η εξής. Ποια είναι τα εμπόδια τα οποία θα πρέπει να αναιρεθούν στον τομέα των υπηρεσιών κυρίως, έτσι ώστε να πετύχουμε τα προσδοκόμενα κέρδη. Τι διορθώσεις έχουμε κάνει μέσω της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Χρειάζεται μια νέα οδηγία ή απλά να εφαρμόσουμε με καλύτερο τρόπο την ισχύουσα. Merci, Madame Ευχαριστώ, euh, l'importance euh, du, du travail Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την τεράστια προσπάθεια που κάνατε. Έχω την αίσθηση ότι στα πλαίσια αυτής της μελέτης έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για τα πιθανά κέρδη ε, της εμβάθυνσης της, ε, της ενιαίας αγοράς. Αυτό είναι και μια προσδοκία των πολιτών μας το να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά που να μην παρουσιάζεται μόνο σαν κάτι το οποίο προκαλεί κέρδη. Δεν θα πούμε το αντίθετο εμείς, αλλά κάθε νόμισμα έχει και την πίσω πλευρά. Υπάρχουν εσωτερικές πλευρές αρνητικές για την εσωτερική αγορά ε, κάποιες περιπτώσεις που δεν είναι στον βασικό στόχος του νομοθέτη, ε, σαν παραδείγμα ο μηχανισμός ε, φορολογικής εναρμόνισης. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν αντιτιθέμενοι στόχοι. Υπάρχουν κάποιες μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ακριβώς αυτήν την ανταγωνιστική μορφή επιδίωξης φορολογίας, πραγματικό άθλημα. Έχουμε λοιπόν από τη μία την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, αλλά η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δείχνει ότι έχει υπάρξει και στρεβλή χρήση του κέρδους αυτού, των δυνατοτήτων αυτών της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, με σκοπό μ, κάποιες ε, συμβάσεις ε, ομαδικές να τις παρουσιάζουν οι εταιρείες αυτές σαν ατομικές συμβάσεις ιδιαίτερα στη Γαλλία γίνεται αυτό. Επίσης το ίδιο γίνεται και για τις online συναλλαγές. Δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις αρνητικές γιατί έχουμε ε, κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με την εγκληματική χρήση ε, κάποιων θεμάτων που άπτονται του αθλητισμού δεν έχουμε δηλαδή μία ποσοστοποίηση κάποιων εσωτερικών χαρακτηριστικών της εσωτερικής αγοράς ή τουλάχιστον έτσι το βλέπουν οι συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πρόεδρε, ο κύριος Ντάν. Να πω προς την κυρία Λάγκεν, από ό,τι νομίζουμε εμείς ε, τα ποσά στα οποία αναφερόμαστε είναι σε αιτήσια βάση. Αλλά μιλάμε για εκτιμήσεις κυρίως τώρα για την οδηγία για τις υπηρεσίες για τον κύριο Στέφανιτς. Ε, το θέμα της εφαρμογής έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως επίσης και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η εξαίρεση κάποιων τομέων από ε, την οδηγία. Υπάρχουν πολλά που πρέπει εδώ να συνεχιστεί, ε, προς τα οποία πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια. Αν μας ζητήσετε να εμβαθύνουμε στα θέματα που αναφέρατε κυρία Ροζιέρ, γιατί όχι. Δεν ξέρω, ίσως να δώσω το λόγο στον Τζάκι για τις για την εφαρμογή της οδηγίας δεν έχουμε νέα στοιχεία και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει νομίζω και σας. Υπάρχει μια πολύ λεπτομερής, έκθεση από το 2011 η οποία διεξήχθη μέχρι τα μέσα του 2012 αφορά τους επαγγελματίες και κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα όπως νομικές υποχρεώσεις κτλ. Το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να δώσει την αυτονομία, την διακανονιστική στα κράτη-μέλη και από την άλλη να μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη-μέλη αυτά για τη μη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. Εν πάση περιπτώσει η οδηγία αυτή εφαρμόζεται με κάπως μέτριο τρόπο θα λέγαμε από τα κράτη-μέλη αλλά δεν υπάρχει αυτή η καταστροφή την οποία πολύ εύκολα διαδίδουν οι εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια λεπτομερέστατη έρευνα της κατάστασης όπως το κάναμε σε επίπεδο λεπτομέρειας το 11 ή μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει ή να το κάνετε όπως έγινε το 2011 μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη δηλαδή να ελέγχει το ένα το άλλο. Διερέθηκαν σε 4-5 ομάδες 4-5 κρατών μελών και ε, υπήρξε ένας αυτοέλεγχος θα έλεγα. Αυτό είχε φανταστικές επιπτώσεις. Ένα κράτος μέλος που έχει ας πούμε μια μικρή νομοθετική ρύθμιση, βλέπει ένα άλλο κράτος που έχει μια βαρύτερη νομοθετική ρύθμιση και λέει γιατί την κάνετε αυτήν, εμείς δεν τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, βλέπετε ότι πολύ καλύτερα γίνεται έτσι το πράγμα από ότι θα μπορούσε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν τα στοιχεία γνωστοποιηθούν, η Επιτροπή σας θα μπορούσε να προσφέρει πολλά. Να μπορούμε να ελέγξουμε ο ένας τον άλλο δηλαδή παρόλα αυτά θα υπάρξει μια κάποια ετερογένεια στα θέματα αυτά και ε, να πω για τις συμβάσεις όπως είπε και ο Τζον Ντάν κάτι. Στις Ηνωμένε Πολιτείες πολύ λιγότερο από την Ευρώπη συνδέεται το ομοσπονδιακό επίπεδο και το πολιτιακό επίπεδο. Οι πολιτείες κάνουν πράγματα χωρίς να ενημερώνουν καθόλου την ομοσπονδία και εμείς εδώ έχουμε το αντίθετο. Τα κράτη-μέλη μπορούν όμως να κάνουν πράγματα χωρίς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βελτιώνοντας την εσωτερική αγορά. Πώς το κάνουν αυτό στις Ηνωμένες Είναι περίπλοκο το θέμα, αλλά μπορούμε να δούμε κάποια βασικά. υπάρχουν επιμέρους διμερείς συμβάσεις ανάμεσα σε ε, πολιτείες για χιλιάδες θέματα στα οποία το ομοσπονδιακό επίπεδο είτε δεν μπορεί να παρέμβει είτε δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει και η κατάσταση βελτιώνεται εδώ. Ίσως αυτός να ήταν ένας τρόπος ε, αντιμετώπισης της διακανονιστικής ετερογένειας. Νομίζω ότι είναι κάτι το πάρα πολύ ε, καλό για την επιχειρηματικότητα να λέμε ότι θα κρατάμε το δικαίωμα νομοθετικής ρύθμισης και παρέμβασης αλλά ίσως θα μπορούσε να δημιουργηθεί ανάμεσα σε λίγες χώρες η συμμαχία των γενναίων που θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε επιμέρους δικές τους βελτιώσεις. Ένα τελικό ε, σημείο, δεν θα μιλήσω εδώ για τους υπόλοιπους συναδέλφους, αλλά στρέψαμε ιδιαίτερο στην προσοχή μας στις 30 σελίδες βέβαια που είχαμε για την αγορά των υπηρεσιών. Δεν είναι ένας αγώνας προς τα κάτω όπως άφησε να εννοηθεί, μάλλον δεν άφησε να εννοηθεί η Γαλλίδα συνάδελφος, αλλά είπε ότι υπάρχουν κίνδυνοι ως προς αυτό. Πράγματι είναι μία δυνατότητα, αλλά η δυνατότητα αυτή δεν έχει επαληθευτεί μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι η χρήση της οδηγίας δεν είναι η σωστή, εκτός όμως από το θέμα της, ε, των ρυθμίσεων για τις διαμεθοριακές υπηρεσίες. Εκεί τα θέματα είναι κοινωνικά εύθραυστα και εκεί η Κοινωνική Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάντως νομίζω ότι δεν είναι σωστό να υποτιμήσουμε την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Αντίθετα έχει δουλέψει αρκετά καλά και μπορεί να προστατεύσει από καταστάσεις όπως αυτή στην οποία αναφερθήκατε. Είναι και άλλα τα θέματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς να αφαιρέσουμε τα φορολογικά δικαιώματα ε, των ε, κρατών μελών των εθνικών διοικήσεων ε, τουλάχιστον να μην θίξουμε το επίπεδο επιβολής στην αυτονομία του. Επομένως χρειαζόμαστε περισσότερα σε αξιολογήσεις ομοτήμων. Για να προσθέσω και εγώ μια παρατήρηση. Λοιπόν, επόμενοι πέντε ομιλητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Ποσφίσιλ. Ένα σύντομο ερώτημα γιατί περνάει και η ώρα. Από τη συζήτηση φάνηκε πολύ καλά ότι με τη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς συνδέεται άμεσα το ζήτημα της εφαρμογής νομοθεσίας. Εγώ στην Τσεχία έχω ευρή εμπειρία με αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ιδιωτικού δικαίου και θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Υπάρχει ποιότητα της εφαρμογής αλλά, του νόμου, αλλά υπάρχει και η εύρυθμη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Κάτι εντελώς διαφορετικό. Και φαίνεται ότι ιδίω στις χώρες που ε, προσχώρησαν τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, και εδώ μιλάμε για τη διάρκεια της ε, δικαστικής διαδικασίας, θα ήταν καλό στο μέλλον να αναλύσουμε πόσο παίρνει η εκδίκαση συγκεκριμένων αντιδικιών ε, στα επιμέρους ε, κράτη-μέλη και ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κουόγκα. Ναι, άκουσα αυτό που είπατε για τον τζόγο στο διαδίκτυο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Υπάρχει και τελευταία νομοθεσία και το Εμνοβασίλειο Βασίλειο ρύθμισε την αγορά, γιατί παλαιότερα το Γιβραλτάρ ε, ρύθμισε την αγορά του το και έπαιρνε όλα τα φορολογικά έσοδα, εκατοντάδε δι ευρώ και τώρα επιτέλου. Δόξα τω Θεώ αποφάσισαν να το ρυθμίσουν. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε αν μπορείτε να εκτιμήσετε το μέγεθος αυτής της αγοράς και τι μπορούν να κάνουν οι ευρωπαϊκές αρχές για να υπάρξει κάποια αναρμόνιση, να γίνουμε ε, μια νέα αγορά. Γιατί στη Γαλλία αποφάσισε να ε, φορολογήσει στον κύκλο εργασιών και να κλείσει την αγορά. Η Εστονία έκανε το αντίθετο. Αφήνει τους πάντες να παίζουν και ε, φορολογεί με ένα 5%. Και η Μάλτα έχει λάβει μέτρα. Η Μάλτα πώς μπορεί να ρυθμίζει την αγορά για την Τσεχία, για άλλους. Πώς διασφαλίζεται έτσι η προστασία των καταναλωτών. Πώς παίρνουν έσοδα από άλλα κράτη-μέλη μέσω του φορολογικού dumping, γιατί περί αυτού πρόκειται. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, είναι βέβαια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν το Γιβραλτάρ έχει μια πολιτική μηδενική φορολόγηση για κάποιου, παίρνει όλα τα έσοδα θα κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εναρμόνιση τη αγορά. Εσεί τι θα κάνετε, θα μα δώσετε καμία συγκεκριμένη πρόταση ή απλά θα συνεχίσουμε στο έλεος ε, των ε, λόμπι. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο, Πρόεδρε, κύριο Σόλτες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ε, προετοίμασαν αυτές τις μελέτες. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει ένα θεματικό τομέα που είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και στα αγαθά και στις υπηρεσίες. Και αναφέρομαι στις δημόσιες προμήθειες. Προσπαθούμε από το 1990 να επεξεργαστούμε ρυθμίσεις για αυτό το τομέα, οι οποίες ακόμα και σήμερα όμως μένουν ανεπαρκείς. Υπάρχουν ε, αρχές τι πρέπει να ε, τηρήσουμε, η τυπικότητα, η διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική. Και εδώ δεν εννοώ διαφάνεια, δηλαδή να έχουμε τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού ε, σε επίσημη εφημερίδα. Όχι. Μιλώ για διαφανή κριτήρια. Εκεί επισέρχεται η διαφθορά. Δεν υπάρχει έλεγχος. Βλέπουμε πολλά παραρτήματα, αυξάνονται, αυξάνεται το κοστολόγιο, το σύστημα φαίνεται ότι δεν λειτουργεί καλά. και θεωρώ ότι είναι ένας ε, τομέας με πολύ ψηλό κίνδυνο διαφθοράς. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε πλήρη αντιστροφή στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Παρόλες τις οδηγίες και τις ε, νομοθετικές πράξεις που έχουμε υιοθετήσει μέχρι τώρα δεν είναι μόνο οικονομική κατηγορία. Οι δημόσιες προμήθειες θα έπρεπε να αποτελέσει ε, κινητήριο μοχλό για τροποποιήσεις σε άλλους τομείς, όπως οι δημοκρατικές ελευθερίες. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη εάν μέσω ενός διαγωνισμού, για παράδειγμα, πετύχαμε τον αρχικό μας σκοπό. Δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπός οι διαγωνισμοί, οι δημόσιες προμήθειες. Θα πρέπει να αποτελέσουν μέσο για την επίτευξη των σκοπών που θέτουμε όταν αποφασίζουμε να κάνουμε έναν τέτοιο διαγωνισμό. Και μετά λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πρέπει να αξιολογούμε κατά πόσο επετεύχθη ο στόχος μας. Επιπλέον, αν η Ευρώπη θέλει να αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, θα πρέπει να διασφαλίσει ένα επίπεδο ελέγχου ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω και το εξής ερώτημα. Εσείς Πώς βρήκατε, πώς καταλήξατε σε αυτά τα στοιχεία για την εξοικονόμηση πόρων στις υπηρεσίες και στα εμπορεύματα. Νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στην νομοθεσία. Για παράδειγμα, για τον ιατρικό εξοπλισμό, για τα συστήματα πληροφορικής και στον τομέα των κατασκευών οι δείκτες που χρησιμοποιείτε στις μελέτες σας είναι χρήσιμοι. Μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να δούμε αν ήταν επιτυχής οι διαγωνισμοί ή όχι. Θα πρέπει να στραφούμε περισσότερο προς την αξιολόγηση με την βοήθεια αυτών των δικτών. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση για την ίδια τη μελέτη. Εντάξει, μπορούμε να εξετάσουμε κατά επιμέρους μέτρα. Το πιο σημαντικό εδώ είναι να μας πούν και άλλοι φορείς, άλλα θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα, για τα συμπεράσματα, για αυτά τα μακροοικονομικά στοιχεία. Γιατί είναι τεράστια τα ποσά. Και τόσο ωφέλη που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε για τους πολίτες μας. Και επί της διαδικασίας λοιπόν υπάρχουν δεκάδες μελέτες, εκθέσεις ερευνητών, αλλά αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη εξαιρετική μελέτη, ιδίω αυτή τη στιγμή. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την εσωτερική αγορά και, την, ε, και το ψηφιακό θεματολόγιο. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν είναι μια μελέτη στο σωρό ή αν εμείς εδώ στην Επιτροπή μας Τη ζητήσαμε, τη θεωρούμε πολύ σημαντική και θα αποτελέσει και βάση για το μελλοντικό μας έργο και ακόμα και το διοργανικό έργο. Μας ε, κατευθύνει προς ε, τα προβλήματα αλλά και προς τις ε, δυνατότητες που έχουμε στους επιμέρους κλάδους. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η μελέτη, αλλά αν τις δώσουμε τη σημασία που δίνουμε στις εκατοντάδες μελέτες που εκπονούνται κάθε χρόνο, τότε τι νόημα έχει η όλη διαδικασία. Και επιτάχυνση χρειαζόμαστε. Εντάξει, καλή εμβάθυνση, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. So I've saved the last question. Τελευταία ερώτηση από μένα. Ήταν εντυπωσιακέ οι εκθέσεις, ιδίω για τα αριθμητικά στοιχεία που είναι μεγάλα ποσά και καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει κάποια πανάκια που θα οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Και όσο πιο πολύ πιέζουμε, τόσο πιο δύσκολο είναι να μπορέσουμε να αποκομίσουμε αυτά τα ωφέλη. Θα ήθελα να σας παροτρύνω να δείτε τις λεπτομέρειες αυτών των εκθέσεων, γιατί οι παρουσιάσεις μονάχα ψάβουν την επιφάνεια. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να βρείτε στις εκθέσεις. Αν θέλουμε να πετύχουμε λοιπόν αυτές τις μεγάλες εξοικονομήσεις, θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες για τις μεμονωμένες δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε και εγώ θα ήθελα να κοιτάξουμε πιο εστιασμένα μεμονωμένες περιπτώσεις και να υπάρξει και μία έρευνα ομοτήμων ε, για τις ε, μελέτες αυτές. Για τις συγκεκριμένες τώρα δράσεις. Εμένα με ενδιαφέρε <clears throat> ιδιαίτερα το όφελος που μπορεί να προκύψει από την άρση των εμποδίων για τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Τι είδου εμπόδια υπάρχουν για αυτές τις επενδύσεις λεγόμενες FDI. Γιατί οι επενδύσεις είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για μας για να μπορούμε να έχουμε την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Αν έχετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα στον τομέα αυτό θα ήθελα να τα ακούσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια και θα δώσω το λόγο πάλι στους εμπειρογνώμονες. Είναι ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα που είπατε. Είναι ενδιαφέρον τα ερωτήματα. το θέμα των, ε, της εφαρμογής τονιστεί σε πολλά ερωτήματα. Είπα ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο μια συνοπτική έκθεση και ήταν τα αποτελέσματά μας ε, κάπως ε, οικοτολογικού χαρακτήρα. Δεν συνδέονται όλα αυτά λοιπόν πλήρως με τη, τα στοιχεία που ερευνάμε. <clears throat> Ίσως θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βάση στην εφαρμογή και να έχουμε καλύτερο έλεγχο των κινδύνων και εφαρμογή κυρώσεων. Ξέρω ότι η Επιτροπή σας έχει εργαστεί πάρα πολύ για τα θέματα ασφάλειας προϊόντων και για την εποπτεία των αγορών ώστε να μπορούν να είναι πραγματικά αποτελεσματικές και αποτελεσματικές σε σχέση με το κόστος για το, τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και αυτό ξέρω ότι σας έχει απασχολήσει στο παρελθόν για την διαδικασία φυσικά να πρόκειται σε εσά να κάνετε μια έκθεση νομοθετική πρωτοβουλίας βάσει του άρθρου 225 εφόσον το επιθυμείτε για την προστασία των καταναλωτών αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση που εναπόκειται σε εσά. Και το σύστημα αμοιβαίας ε, αξιολόγησης, η αξιολόγηση από μοτίμους όπως είπε η πρόεδρος, είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται στην ε, νομοθετική δραστηριότητα. Ήταν ό,τι αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η διαδικασία. Υπάρχει και μια μεγάλη μελέτη που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία παραπέμπουμε κι εμείς. <clears throat> Ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον πρόεδρο Μπαρόζο, νομίζω τον Νοέμβριο του 2010, και ζητήθηκε από την Κομισιόν να εκπονήσει μια έκθεση για το κόστος της μη Ευρώπης ουσιαστικά. Η έκθεση αυτή ε, βγήκε χωρίς ε, βάια και κλάδους πέρσι, αλλά δεν έχει αναφερθεί πολύ, δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι μια ευρεία, ε, ευρέως πεδίου μελέτη και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να κάνει περισσότερα στους τομείς που ανέφερε ο Τζεφ προηγουμένως στο λιανεμπόριο. Ξέρω ότι το έχετε ζητήσει εσείς ως Επιτροπή αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις που μπορεί να βελτιωθεί <clears throat> η κατάσταση για το λιανεμπόριο και την, ε, τα θέματα επιμελητίας για την παράδοση προϊόντων. Και το Ίδρυμά μου, το EPRS, είναι έτοιμο πάντα να υποστηρίξει ό,τι θέλετε να κάνετε σε σχέση με ακροάσεις ή συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα. Μπορώ να δώσω λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους. Ένα μοναχά. σημείο για αυτά τα οποία μας είπαν οι δύο ε, ευρωβουλευτές για την, την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Το θέμα της επιβολής αυτών των ρυθμίσεων είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει με τον προηγούμενο πρόεδρο της Επιτροπής σας επανειλημμένα. Είχαμε λοιπόν συζητήσει αναλυτικά και στον τομέα των δημοσίων ε, ε, προμηθειών είχαν, είχαν υπάρξει κάποιες λύσεις. Οι θεσμοί των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για την διόρθωση των προβλημάτων ε, αυτό το προβλέπει και η κοινοτική νομοθεσία. Επανειλημμένα εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε ε, τα συστήματα αποκατάστασης τα εθνικά Ξέρετε ότι η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Ήδη ε, μέχρι το 12 είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο δεν λειτουργεί το σύστημα και υπάρχουν γιγαντιαίες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, στα πλαίσια της λειτουργίας ή της μη λειτουργίας του συστήματος και τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να κάνουν τίποτα γύρω από αυτό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Είναι τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης, ε, ε, ίσως και θέματα διαφθοράς, αλλά μία βελτίωση σε επίπεδο επιβολής θα προκαλέσει πάρα πολλές δυσκολίες με τα κράτη-μέλη, αλλά ίσως και να αξίζει τον κόπο να την επιδιώξετε. Εσείς θα το αποφασίσετε. Το πρώτο βασικό θέμα αφορά τις απάτες και την διαφθορά. Υπήρξε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ο τομέας των δημοσίων προμηθειών ήταν κατεξοχήν προς εξέταση. Είναι μια πραγματική ανησυχία γιατί επηρεάζει πάρα πολύ την κατάσταση. Κάποιες πρακτικές αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 με 25% των συμβάσεων και αυτό είναι μια τεράστια ανησυχία. Και υπάρχει ένα τμήμα της έκθεσής μας το οποίο αναφέρεται στις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης σχετικά με τα δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο τα συλλέξαμε. Εμείς πήραμε στοιχεία πρώτον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει κάποιες εκτιμήσεις γύρω από το σύνολο ε, των ε, συμβάσεων και ε, έχει και τις τελικές αξίες, το τι πληρώθηκε ακριβώς και γενικά έτσι μπορέσαμε να πάρουμε κάποια στοιχεία προς ενημέρωση. προσπαθήσαμε να δούμε τις διαφορές ανάμεσα σε αυτό το οποίο πίστευαν ότι θα πληρωθεί και σε αυτό το οποίο τελικά πληρώθηκε. Ίσως τελικά κάποια μία έλλειψη, αδυναμία μάλλον εξοικονόμησης χρημάτων οφείλεται και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η συγκεκριμένη οδηγία, οι συγκεκριμένες οδηγίες. Ένα άλλο σημείο τώρα αφορά στο αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά για να εκτιμήσουμε ε, την επιτυχία ή όχι συνολικά της προσπάθειας. θα προσπαθήσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τον πιο δυνατά αναλυτικό τρόπο, να δούμε τι εξοικονόμηση πιστώσεων έχει υπάρξει και επί τη βάση αυτών των διαπιστώσεων και υποθέσεων να εκτιμήσουμε ε, την δυνητική, ε, το δυνητικό κέρδος. Αλλά θα πρέπει εμείς να κατανοήσουμε πρώτα το τι δούλεψε. Ευχαριστώ. για τις επενδύσεις είχαμε κάποιους περιορισμούς σε σχέση με τα δεδομένα τα οποία πήραμε από τον ΩΣΑ που συλλέγει τα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δεν μπαίνουν σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας και για τα FTI που προκαλούνται μερικές φορές στο διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζουν τις χώρες ή οι διεθνείς επενδυτές και αυτό είναι αν θέλετε και μία από τις βασικές προειδοποιήσεις που μας δείχνει η έκθεση αυτή. Λέμε ότι υπάρχει πιθανό κέρδος από τη μείωση αυτών των εμποδίων, αλλά απαιτείται έρευνα μεγαλύτερη και περισσότερη για να δούμε ακριβώς ποιος είναι ο λόγος που τα δημιουργεί. Λοιπόν, ξέρουμε βέβαια εμείς ποια είναι τα στοιχεία, δεν μπορούμε όμως να τα εντοπίσουμε με τον πιο καλό τρόπο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι μας δώσατε πάρα πολύ υλικό και πάρα πολύ ψηλά ποσά εφόσον τα πετύχουμε βέβαια. Ευχαριστώ. then going to move on to our next item of business because we're running a little bit short. Um, this is the report. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ας περάσουμε λοιπόν ε, στην ε, έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ο Σέρτζο Καχαράτη είναι εισηγητής. Θα σχόλια στις τροπολογίες. Θα υπάρξει μία ανταλλαγή απόψεων. Θα καλήσω πρώτα τους σκιώδεις να πάρουν τον λόγο. Να σας θυμίσω ότι θα ψηφίσουμε τις 58 τροπολογίες αύριο. Έχουμε τέσσερις συμβαστικές Και από ό,τι... Ή μάλλον να ευχαριστήσω όσους ε, εργάστηκαν με τόσο ταχύ τρόπο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ τροπολογίε τόσο σύντομα. Ελπίζουμε αύριο να εγκρίνουμε την ε, γνωμοδότηση γιατί ε, στην Ήμικο θα ψηφίσουμε στις 7 Το Οκτωβρίου και θα περάσουμε στην Ολομέλεια στα τέλη Οκτωβρίου. Σέργιο, να σου δώσουμε το λόγο για μερικά λεπτά. Ένα λεπτό κάθε ε, σκιώδης. Grazie. Κύριο Σκοφεράτη, ευχαριστώ κάποια πρώτα λόγια για τους συναδέλφους οι οποίοι είναι καινούργοι στην Επιτροπή για να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο μέσα στο οποίο ε, εξετάζουμε τη συγκεκριμένη έκθεση. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδιαίτερα στην αρχική του φάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, παράγει τρεις εκθέσεις. Η μία είναι της Επιτροπής ΕΚΟΝ και αφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία Μία άλλη είναι της απασχόλησης που αφορά τα θέματα της απασχόλησης και μετά είναι η δική μας που αναφέρεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Όταν κλείνει ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως γίνεται αυτό σήμερα, ε, προετοιμάζεται μία άλλη έκθεση, όπως μας θύμισε η Βίκη, που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες και οι άλλες επιτροπές παρουσιάζουν και αυτές μία γνωμοδότηση η οποία σχολιάζει το στάδιο προόδου ε, του εξαμήνου. Συμβατικά τώρα ποιος, όποιος κάνει την αρχική έκθεση είναι και τελικός γνωμοδότης. Οι χρόνοι που προβλέπονται είναι πάρα πολύ μικροί, υπάρχει επιταχυμένη διαδικασία και έτσι γι' αυτό αύριο θα κληθούμε να ψηφίσουμε. Προσπαθήσαμε μέσα από το κείμενο αυτό, σε συνεργασία με τους συναδέλφους, τους οποίους ευχαριστώ, να ενισχύσουμε την ιδέα ε, του ρόλου του Κοινοβουλίου στην εσωτερική αγορά και το πού μπορεί η εσωτερική αγορά να διασταυρώνεται με τις οικονομικές πολιτικές. Λάβαμε υπόψη μας την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα για το κομμάτι το οποίο αφορά τις συστάσεις ανά χώρα. Έχουν υπάρξει κάποια βήματα προόδου, υπάρχουν πολλά τα οποία μένει να γίνουν, αλλά θα τα εξετάσουμε αυτά στα πλαίσια ε, του χρόνου που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τις ανησυχίες που έχουμε εκφράσει και για τις ελλείψεις συνεργασίας στο φορολογικό κομμάτι και για τον εξυγχρονισμό των δημόσιων διοικήσεων. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα εμείς να θεωρήσουμε την εσωτερική αγορά σαν τον τρίτο πυλώνα, κάτι το οποίο για μας είναι δεδομένο, αλλά για το σύνολο του Κοινοβουλίου δεν έχει ακόμα γίνει αντιληπτό και στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 η οποία έχει κλονιστεί βαρύτατα από την κρίση Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και το ρόλο των δημοσίων επενδύσεων, ιδιαίτερα σε ορισμένους κομβικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η έρευνα και η καινοτομία. Είναι μεγάλη επίσης ανάγκη υψηλού επίπεδου ποιοτικού δημοσίων υπηρεσιών μέσω του εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και μέσω της δημιουργίας της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, ένα από τα βασικά θέματα των επομένων μηνών. Είναι 58 όπως είπα οι τροπολογίες που κατετέθησαν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους οι οποίοι ε, έχουν συντάξει τις τροπολογίες αυτές οι οποίες όλες εντάσσονται στο πνεύμα και την λογική που προανέφερα. Κάτι τέτοιο λοιπόν έρχεται αρρωγός στην δική μας προσπάθεια. Εγώ ίδιος με τους συναδέλφους μου χρειάστηκε να καταθέσουμε τέσσερις συμβιβαστικές τροπολογίες σε κάποιες από αυτές υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές τις οποίες ελπίζω να καλύψουμε το μεσημέρι έτσι ώστε αύριο στην ψηφοφορία να καταθέσουμε τις τροπολογίες τις οποίες εν πολλής θα συμμεριζόμεθα. Οι τροπολογίες αυτές ή μάλλον οι συμβιβαστικές τροπολογίες ακριβώς καλύπτουν τις συστάσεις αναχώρα πρώτον, την ανάγκη δημοσίων επενδύσεων για την πραγματική οικονομία, τον ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών για την κοινωνική συνοχή και το θέμα του εξυγχρονισμού των δημοσίων ε, διοικήσεων. Σας ευχαριστώ που συνεισφέρατε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα το κλείσουμε το θέμα αυτό. Όπως είπα είμαστε σε μια φάση πολύ προχωρημένη. Ελπίζω αύριο να κλείσουμε το δικό μας ίτερ, τη δική μας διαδικασία. Με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ή κάποια επιμέρους στοιχεία. Ε, μπορώ να σας τα δώσω στην απάντησή μου σε ερωτήσεις σας. Um, e- Ευχαριστώ. Από το Έλκο Κάπρος, ή Λίκο Κάπρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κομφέρατη για το έργο του, πρώτα απ' όλα. 58 τροπολογίες έχουν κατατεθεί και 4 συμβιβαστικού χαρακτήρα τροπολογίες, μέσω των οποίων μπορεί να βελτιωθεί το κείμενο. Πιστεύω ότι η συνεργασία ήταν πολύ καλή με τον εισηγητή και τους συνεργάτες του. Εδώ υπάρχει ένα σημείο εκκίνησης για την έκθεση αυτή που διατρέχει και όλη την έκθεση και που έχει ακριβώς σαν στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Η, το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στην ε, εσωτερική αγορά είναι πολύμορφο και πολυσχηδές. Αυτό αποτελεί πρόβλημα, πολλές φορές εμποδίζει την ε, ε, περάτωση της εσωτερικής αγοράς είναι κάτι το οποίο εκρεμεί ακόμα και αυτό εγκυμονεί προβλήματα. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτών των ρυθμίσεων επίσης είναι ένα περαιτέρω πρόβλημα γιατί και πάλι λόγω της μη αποτελεσματικής εφαρμογής δεν μπορούμε να επιτύχουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε και φυσικά υπάρχουν και μεθοδολογικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κομφεράτη ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ένα κέριο σημείο και είναι η ελπίδα όλων μας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να είναι ο κινητήρας της ανάπτυξης της οικονομίας μας και πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό απασχόλησης, να τονίσουμε το ρόλο της καινοτομία και να εξασφαλίσουμε και την κοινωνική ε, ενσωμάτωση. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε εναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης υποστήριξη και υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στο προηγούμενο σημείο όπου οι εμπειρογνώμονες μας εξήγησαν ότι είναι απαραίτητη μια κάποια φορολογική εναρμόνιση για να έχουμε <clears throat> τα μεγαλύτερα ωφέλη. Εγώ πιστεύω όμως ότι δεν χρειαζόμαστε τόσο μια φορολογική εναρμόνιση, αλλά καλύτερα περισσότερη ενημέρωση, αμοιβαία ενημέρωση για το τι πράττουν τα διάφορα κράτη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα φοροδιαφυγής ή για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν την αύξηση ή μείωση των φορολογικών συντελεστών. Αυτό θα μου φαινόταν, λοιπόν πάρα πολύ χρήσιμο για τι τέσσερι τώρα συμβαστικέ τροπολογίες. Πιστεύω ότι σε γενικέ γραμμές καλύπτουν τι τροπολογίε, οι οποίε έχουν κατατεθεί, επομένω μπορούν να τύχουν υποστήριξη από εμά. Εγώ έχω τώρα δύο προτάσει για τι οποίε έχω ήδη συζητήσει με τον κύριο Κομφεράτη για τις συμβαστικές τροπολογίες 2 αλλά και 3 για την υπαριθμόν 2 πρόκειται για τις λεγόμενες νέες πηγές, τις νοπές πηγές, όπως λέγεται. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διαγραφεί αυτή η διατύπωση, γιατί εδώ δεν πρόκειται για μια ορολογία η οποία είναι δόκιμη στον οικονομικό τομέα. Έχω ένα πρόβλημα λοιπόν με αυτή την ορολογία. Για την τροπολογία τώρα 3, και εδώ θα ήθελα να διαγράψουμε μια λέξη. Γενικά συμφωνώ με την συμβιβαστική ε, τροπολογία, με την κατεύθυνσή της, αλλά η πλήρης εξάλληψη της ένδυας είναι ένας μακρόπνος στόχος και δεν μπορούμε να τον επιτύχουμε εύκολα. έχει αναφερθεί το θέμα της Ένδειας και πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο στόχος η πλήρης εξάλληψης της ε, Ένδειας. Μπορούμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτός ο στόχος είναι δύσκολο να επιτευχθεί και γι' αυτό δεν πρέπει να αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε αυτό το κείμενο, όπου δεν είναι και το κύριο θέμα. Αυτά οι παρατηρήσεις μου και ελπίζω ότι και το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά. Και γενικά η ομάδα μου υποστηρίζει το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Εγώ είμαι ισχυώδης των συντηρητικών. Στον εαυτό μου θα δώσω και το λόγο. Είναι καταρχήν σημαντικό να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι το εξάμεινο, το οικονομικό εξάμεινο δεν αφορά μοναχά την μακροοικονομική, αφορά όλη την οικονομία και η έκθεση, η οποία, μια έκθεση που εξετάζει την εσωτερική αγορά είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί αναλύει και ειδικά στοιχεία της ε, ενιαίας αγοράς και αυτό έχω καταθέσει και κάποιες τροπολογίες σε σχέση με τα δίκτυα, με τις υπηρεσίες, την ψηφιακή οικονομία και εκεί μπορούμε να είμαστε ίσως και πιο συγκεκριμένοι και αυτό το στόχο έχουν οι τροπολογίες μου. Συμφωνώ με τον εισηγητή για την ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκής υποστήριξη για τους πολίτες και τις ε, επιχειρήσεις όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της εσωτερικής αγοράς. Μπορεί να υπάρξει λοιπόν και κάποια μνήα στην για την καλύτερη χρησιμοποίηση αυτών των ευκαιριών που παρέχει η αγορά, παραδείγματο χάρη στον χώρο των συμβάσεων. Το να εξασφαλίσουμε επίσης ότι υπάρχει επαρκής υποστήριξη για τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόσουν την νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η εκπόνηση αυτής της νομοθεσίας, θα θέλουμε τα κατημέρια ή δυνατόν να την εφαρμόσουν με το σωστό τρόπο και να επιτυγχάνουν τους προσδοκόμενους στόχους. Και αυτά που συζητήσαμε για τους εμπειρογνώμονες μας σήμερα το πρωί, είτε μέσα από το εξάμεινο, είτε με συνεργασία χωρών, όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά στη νομοθεσία μας, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. Πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν και σημαντικά είναι τα, και το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις. Μας είπαν το πρωί ότι υπήρχαν μεγάλα εμπόδια για τις επενδύσεις, ιδίως τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και η πρόσβαση σε ε, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και για μεγάλα σχέδια. Και υποστηρίζω πλήρω τον τελευταίο ομιλητή, την τελευταία ομιλήτρια μάλλον για αυτά που είπε για τα νοπά χρήματα, τα καινούργια χρήματα. Γενικά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι η, η έκφραση αυτή δεν μου φαίνεται πολύ, μου φαίνεται λίγο παράξενη από την, ε, από την οικονομική σκοπιά. Ίσως θα έπρεπε να βγει αυτή η λέξη από την ε, συμβαστική τροπολογία και σας ευχαριστώ για τις συμβαστικές τροπολογίες πως βλέπω σε περαιτέρω συζήτηση προτού φτάσουμε στην ψηφοφορία. Αλλά σίγουρα ξέρουμε όλοι ότι έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Ήμουν και εγώ μία από τις εισηγήτριες για την οικονομική διακυβέρνηση που οδήγησε στο Ευρωπαϊκό εξάμεινο, δεν χρειαζόμαστε μονάχα τις μακροοικονομικές ε, αναλύσεις, αλλά πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και σε σχέση με την συνολική οικονομία. Και μας βοηθάει το να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Από τους φιλελεύθερους κ. Γκόλτζετ. Μπορείτε να μου Είστε πώς... Γκόλτα. Εύκολο, εύκολο. λοιπόν, άμα το συνηθίσει θα το λέτε πιο εύκολο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Πρόκειται για μια πολύ καλή πρόταση και τον ευχαριστώ και για τη συνεργασία του στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι συμφωνούμε και για την παράγραφο 5. Στην αρχή ζητούσαμε ισχυρές πιστώσεις για την ενίσχυση της οικονομίας των κρατών μελών. Ε, φρέσκο χρήμα, ωραία πράγματα αυτά, αλλά δυστυχώς ε, τα όνειρα αυτά δεν βοηθούν και συνήθως οι άμεσες ε, τέτοιες ενέσεις δεν βοηθούν επίσης. Ίσως να καταστήσουν την κρίση ακόμα και χειρότερη. Η ανάκτηση της οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί μόσο. Ε, μόνο μέσω πολιτικών ε, στραμμένων προς το μέλλον και σκληρών αποφάσεων. Ενίσχυση των μικρομεσαίων, πρόσφαση των μικρομεσαίων στη χρηματοδότηση, βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον, αυτά τα οποία πέτυχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα, ναι μεν κρατάει τα επιτόκια χαμηλά, υπάρχει ανταλλαγή ομολόγων ανάμεσα στις χώρες, αλλά δυστυχώς ε, δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων. Δεν υπάρχει δυνατότητα εγγυήσεων των δανείων αυτών. Και αυτό πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να βοηθήσουν την οικονομία και να δώσουν θέσεις εργασίας στους νέους. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στις μικρομεσαίες έτσι ώστε να μπορέσουν να τύχουν πραγματικής στήριξης. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, προβλέπει πιστώσεις προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω να το πετύχουμε. Στήριξη της ψηφιακής οικονομίας, στήριξη του τηλεπικοινωνιακού τομέα, αυξημένη χρήση του e-government. Εγώ δεν είμαι Εσθονός, αλλά δείτε τι γίνεται στην Εσθονία. Ψηφίζουν online στην Εσθονία. Είναι θέμα αποτελεσματικότητας. Αυτό χρειάζεται η Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε στον τομέα αυτό και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σωστά και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Um, Ο κύριος Δεγιόν, ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση ουσιαστικά αντικατοπτρίζει όλη τη δουλειά που έχει γίνει στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, κατά το παρελθόν. Θυμάμαι την, πρωτοβουλία, γνωμοδότηση πρωτοβουλίας ε, του κυρίου Σφαμπ για την εσωτερική αγορά και το ευρωπαϊκό εξάμεινο που ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιες πολιτικές ομάδες θα το πιέσουν, άλλες θα το καταψεφίσουν. Ακόμα και τότε θα είχαμε αυτήν ε, τη διελκυστίδα. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε να μην ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερο το σύνολο της ε, Επιτροπής ε, εσωτερική αγορά να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, γιατί ακόμα είμαστε πολύ σημαντικό κομμάτι των ε, διατάξεων εφαρμογής. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο σημείο που μπορούμε να πούμε να ότι θα υπερψηφίσουμε αύριο. Από πλευράς μου έχω μερικές παρατηρήσεις που θα πρέπει να επιληθούν ε, σήμερα το απόγευμα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι μιλητές, αν επικεντρωθούμε ε, στην κύρια ουσία της μελέτης, της έκθεσης, συγγνώμη, τα πράγματα είναι πιο απλά. Όσο προσθέτουμε στοιχεία, δυσκολεύουν τα πράγματα. Για παράδειγμα, η πρώτη συμβαστική τροπολογία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διατύπωση για τις ε, διαθερωτικές μεταρρυθμίσεις, structural reforms. Είναι μάλλον ασαφής αυτός ο όρος. Μιλάμε για φορολογική μεταρρύθμιση που είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή στη χώρα μου, στις κάτω χώρες ή μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, τι εννοούμε, δεν είναι σαφές και οδηγεί σε μια τέρμονη συζήτηση. Καλό θα ήταν να το διαγράψουμε λοιπόν, να επικεντρωθούμε στην εσωτερική αγορά και έτσι είναι πιο εύκολη η επίτευξη συνένεση στην Επιτροπή μας. Για τη δεύτερη συμβιβαστική Γέλασα τον είδα αυτό το fresh money, τα νοπά τα χρήματα, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι είναι βρώμικο το χρήμα, άλλοι ότι είναι καθαρό. Νοπό όμως δεν το έχουμε ακούσει, εννοούμε ουσιαστικά περισσότερα χρήματα. Βέβαια, τα πιστά χρήματα δεν είναι πάντα η λύση. Συμφωνώ λοιπόν με την Πρόεδρο που είπε να το διαγράψουμε. Έτσι και αλλιώς δεν αφαιρεί κάτι από την έκθεση. Όπως και να έχει, πάντα υπάρχει δυνατότητα ο καθένας να επενδύσει όσα, όσους δημόσιους και δυτικούς πόρους επιθυμεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν για να το αφήσουμε εκτό. Και τέλο, για τι δημόσιε υπηρεσίε, στην τρίτη συμβιβαστική. Και πάλι. Λυπάμαι που αντικαταστήσαμε το high quality με quality. Υψηλή ποιότητα το κάναμε σχέτη ποιότητα, αλλά εντάξει καταλαβαίνω. Μετά για τις ε, προσιτές δημόσιες υπηρεσίες, προσιτές οικονομικά, είναι εξίσου σαφής αυτή η διατύπωση. Το τι είναι προσιτό και τι όχι είναι πολύ υποκειμενικό. Και βγάζουμε το υψηλή ποιότητα δημόσιε υπηρεσίε και προσιτέ δημόσιε υπηρεσίε. δεν βελτιώνει τα πράγματα. Το τελευταίο σημείο, εντάξει, το διαπραγματευόμαστε. Το πιο σημαντικό είναι η πρώτη συμβαστική και αυτό που είπα για τα νοπά χρήματα. Και για το δεύτερη συμβαστική. Αν βρούμε λύση, και πραγματικά το ελπίζω, τότε μπορώ να ήδη να πω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ψηφίσουμε πέρα αύριο. Thank you. Pascal. Ευχαριστώ. Πασκάλ Ντιουάν. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, Πρόεδρε. Thank you. Um, so I... Ευχαριστώ. Ένας ακόμα ομιλητής, η Άννα Μαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Κονφεράτη για την εξαιρετική αυτή γνωμοδότηση. Συμφωνώ με όλους τους προηγούμενους ομιλητές, εκτός από τον κύριο Ντεγιόγκ, το φίλο μου, που γιατί είναι πολύ σαφέ τι είδου μεταρρυθμίσει πρέπει να γίνουν. Η Επιτροπή έχει πει ότι πρέπει να ανοίξει αγορά υπηρεσιών, για παράδειγμα. Ακριβώ σε, σε αυτό το πράγμα αναφερόμαστε. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Σκιώδη από το ΕΛΚ για τις συμβουλευτικές τροπολογίες. Το fresh, όλοι το σχολίασαν ήδη, τι σημαίνει νοπή, φρέσκη πόρη. Ας επικεντρωθούμε στο πραγματικό σκοπό της έκθεσης. Θέλουμε να θέσουμε επικεφαλής της σημερινής διάταξης και στο Κοινοβούλιο και ε, στα κράτη-μέλη ότι η νέα αγορά είναι βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρέπει να συνδεθεί λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με αυτή τη δυνατότητα της ε, αναθεώρησης της στρατηγικής για το 2020. Δεν χρειάζεται να πάμε προς κάθε κατεύθυνση. Πρέπει απλώς να αξιοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε για να επιτύχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Όχι να δώσουμε και άλλους πόρους. Και είναι θετικό που τουλάχιστον έχουμε επικεντρωθεί στην ε, αποτελεσματικότητα, στην αποδοτική χρήση των πόρων, στην καινοτομία, στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στον τομέα των υπηρεσιών. Γιατί εκεί ξέρουμε ότι έχουμε το υψηλότερο, τις μεγαλύτερες δυνατότητες για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Εκεί συντείνουν όλα τα στοιχεία, όλες οι μελέτες μας. Επομένω το Fresh μπορεί να βγει και να επικεντρωθούμε στις δυνατότητες της ε, ενιαίας αγοράς και όχι σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Εντάξει, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα ψηφίσουμε αύριο. Α, ναι. Έχει μείνει κάποιος που θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Η έκθεση η Στρατηγική Ευρώπη 2020 είχε υποσχεθεί τον παράδεισο και στον τομέα της ανάπτυξης και στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης γενικότερα και της απασχόλησης. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Έχει υπάρξει μια πλέον χρόνια ανησυχία, ανασφάλεια και διάψευση των προσδοκιών. Ο κύριος Κοφεράτη και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου προτείνει να λύσει τα προβλήματα αυτά κάνοντας βήματα άκρητα προς τα εμπρός μέσω της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Κάτι το οποίο θα μας πρόξει ακόμα περισσότερο προς τη φτώχεια, την ανέχεια και τη δυστυχία θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ε, ενιαία αγορά, η εναρμονισμένη αυτή αγορά είναι μια ουτοπία και μια οικονομική αποτυχία ταυτόχρονα. Ε, η υπογραφή της Ατλαντικής Συμφωνίας θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις. Η Γαλλία πεθαίνει από τις ε, αποφάσεις αυτές. Το απέδειξαν οι τελευταίες εκλογές, οι ευρωεκλογές. Νομίζω ότι οι Γάλλοι θέλουν πλέον να απορρίψουν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική που προωθεί αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν υπάρχουν ε, ε, κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες. Σήμερα το απόγευμα θα επανεξεταστούν, θα διανεμηθούν σε όλα τα μέλη και στην συνάντηση των συντονιστών το απόγευμα θα συζητήσουμε τα θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Έχουμε κάποια καθυστέρηση λόγω ακριβώς ε, της νεότητας αυτού του Κοινοβουλίου και της ανάγκης προσαρμογής στους νέους ρυθμούς. Αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι η ε, οι τροπολογίες αυτές ε, να μοιράζονται στα μέλη μας με περισσότερο χρόνο. Πάντως όλοι προσπάθησαν και ιδιαίτερα με τόσα νέα μέλη θα πρέπει να, να κυκλοφορούν οι συμβιβαστικές προτάσεις νωρίτερα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ όλους. Τέλος. Uh,